Κυρίες και κύριοι, εάν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φερνάντο Τζεντιλίνη, Θυμίζει Κατενάτσιο και Ιταλία το όνομά σας, ε, κύριε Τζεντιλίνη. Ο κ. Τζεντιλίνη είναι ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαδικασία ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής. Σήμερα το πρωί. Συζητήσαμε σήμερα το πρωί για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, και θα συζητήσουμε στη συνέχεια για τα θέματα των πολέμων αντιπροσώπων και όλα αυτά δείχνουν με ποιο βαθμό, σε ποιο βαθμό μάλλον οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε βίες αντιπαράθεσης στην ε, περιοχή. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή όλα αυτά να δώσουν λαβή σε διαπραγματεύσεις και σε πρόοδο με τη διαδικασία του Όσλο, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε τελικά σε μια αξιόπιστη διαδικασία συζητήσεων που να οδηγήσει σε, ε, ε, σε δύο κράτη, στην, ένα Ισραηλινό κράτος και ένα Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 Κύριε Τζεντιλίνη, λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω από εσά ιδιαίτερα με ποιο τρόπο το κουαρτέτο, η τετραμερής δηλαδή διάσκεψη, εργάζεται για τα θέματα αυτά και πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για νέες διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά της ε, ειρήνευσης στο Παλαιστινιακό. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει επιστροφή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και κάποια πρόοδο στι διαπραγματεύσεις. Και φυσικά εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω τα λίγα λεπτά αυτά για να σας περιγράψω το πώς βλέπω τα πράγματα. Βρίσκομαι εκεί. Εδώ και έξι μήνες είμαι εκεί, στην Ιερουσαλήμ, Συζητώ και με τις δύο πλευρές. Θέλω να πω και αυτό που είπε και είπατε εκπρόσωπος εδώ και 15 μέρες περίπου, να αναφερθώ σε αυτά που μας είπε. Και θα εστιαστώ και στις δραστηριότητε του κουαρτέτου. Είναι σημαντικές, όπως υπενθυμίσατε. Θα αναφερθώ σε τρία στοιχεία, εντάχει. Ένα σημαντικό σημείο είναι να δούμε τι γίνεται επί τόπου πώς θα σταματήσει η βία και τι προσπαθούμε να κάνουμε με τους εταίρους μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά πώς να ξεκινήσει η πολιτική διαδικασία. Και εκεί θα εστιαθώ στη στρατηγική του κουαρτέτου. Να εφαρμόσουμε επιτόπου μέτρα για οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Να δημιουργηθούν συνθήκες για συνομιλίες που θα έχουν νόημα όταν θα είναι κατάλληλη στιγμή. Και μετά συντομία πώς ο πολιτικός ορίζοντας θα είναι ανοιχτό και ποια θα είναι η δίωδος εισόδου για τις συνομιλίες. Να πω εξ αρχής κάτι. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είναι ενεργός φορέας στην προσπάθεια και θέλω να περιγράψω γενικά τι κάνουμε. Οι διάφοροι θεσμικοί φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων ημών με ύψιλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σκληρά, πολύ σκληρά, με τους διεθνείς εταίρους, τη ΣΥΠΑ και άλλα μέλη στο κουαρτέτο για να στηρίξει τις προσπάθειες των ηγετών, να τεθεί τέρμα στη βία και να ξεκινήσει κάποια πολιτική διαδικασία εκ νέου. Το κουαρτέτο ήταν πολύ δραστηριό τον τελευταίο μήνα, συναντηθήκαμε με συναδέλφους επιτόπου και έγινε και μεγάλη σημαντική συνάντηση στη Νέα Υόρκη και μετά στη Βιέννη πριν από 15 μέρες περίπου. Είναι σημαντικό αυτό. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέμειξε τοπικούς εμπλεκομένους φορείς Αίγυπτο, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία στις συνομιλίες διότι πιστεύουμε ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στηρίζοντας τις προσπάθειες των δύο πλευρών έκανα αρκετά ταξίδια στην περιοχή το καλοκαίρι πήγα στο Κάιρο, στο Αμάν, στο Ριάντ και καταλήξαμε στην πρόσκληση του Κουαρτέτου να συναντηθεί με τους περιφερειακούς παράγοντες στη Νέα Υόρκη τέλος Σεπτεμβρίου. Περιφερειακή πολιτική δηλαδή αφορά το θέμα και είναι σημαντικό να αναφερθεί. Πρώτα, η βία. Η κατάσταση είναι, πώς να το πω, αργώς βελτιούμενη στην Ιερουσαλήμ, παραμένει όμως τεταμένη με πολλά επεισόδια στην υπόλοιπη δυτική όχθη, κυρίως κοντά στη Χευρών. Δεν είναι καλή κατάσταση. Η ηρεμία στην Ιερουσαλήμ είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας, των ΙΠΑ, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κέρι που πήγε στο Αμάν πριν από κάποιες εβδομάδες, προσπαθώντας να ηρεμήσει την κατάσταση κοντά στους ε, ιερούς τόπους των ε, Ιεροσολύμων προσπάθεια να παραμείνει καθεστική τάξη και να αναγνωριστεί ο ιδιαίτερος ρόλος που μπορεί να παίξει η Ορδανία. Όλα αυτά συνέβαλαν στον, στην επικράτηση της ηρεμίας, γίνεται προσπάθεια επιτόπου, ούτως ώστε να υπάρχουν καθημερινές διευθετήσεις για την ομαλή εξέλιξη της κατάστασης στους Αγίους Τόπους. Η ΕΠΑ στήριξε, στήριξαν την προσπάθεια και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης εξελίξεις επιτόπου. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να σταματήσει η βία. Και αυτό είναι το βασικό που έχω να πω. Χρειαζόμαστε πολιτική διαδικασία, κάποιο είδους πολιτική διαδικασία επιτόπου, οι δύο να ξεκινήσουν την προσπάθεια για να μειωθεί η βία και στην υπόλοιπη περιοχή, Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους και το κουαρτέτο προσπαθεί να δει αν είναι εφικτό να επανεκκινήσει κάποια προσπάθεια σταδιακή επιτόπου που θα ηρεμήσει την κατάσταση, θα καθησυχάσει τα πράγματα και θα προετοιμάσει από την άλλη και το έδαφος για ε, συνομιλίες οι οποίες θα έχουν νόημα που θα ξεκινήσουν όταν είναι σωστή στιγμή. Οι διεθνείς ηγέτες και είπα ότι εκπρόσωπος περνά το μήνυμα, περνά το μήνυμα ότι είναι τώρα ε, η στιγμή που χρειάζεται ηγεσία και από τις δύο πλευρές. Και αυτό που ζητούμε και ζητήσαμε και ζητά το κουαρτέτο και στην Νέα και στη Βιέννη είναι αλλαγή πολιτικής. Σειρά μέτρων που θα επιφέρουν αλλαγές. Να δοθεί περισσότερη δύναμη στους Παλαιστινίους διαφυλάσσοντας την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να δούμε, αυτό επεξεργαζόμεθα και στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα, και εν τέλει θα ενισχυθεί η λύση των δύο κρατών με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς ίσως διολυστήσει αυτή η λύση. Πολλές συμφωνίες έχουν επιτευχθεί κατά το παρελθόν. Κάποιες από αυτές μπορούν να εφαρμοστούν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν βήματα που μπορούν να εξετάσουν οι δύο πλευρές, οικονομικής φύσεως, θεσμικής φύσεως, υπό τη μορφή μέτρων για την ασφάλεια ε, και όλα αυτά θα έχουν θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τελικά οι δύο πλευρές θα πρέπει να αποφασίσουν. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να γίνει. Για να είμαι ειλικρινής υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ των δύο πλευρών. Το καλό είναι ότι και οι δύο, λένε, οι δύο πλευρές δεν ότι είναι έτοιμες να κινηθούν επί τόπου. Απ' την άλλη υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των Παλαιστινίων και εκείνων που είναι έτοιμοι να πράξουν οι Ζαλινοί. Εμείς είμαστε στη μέση των δύο. Τώρα δοκιμάζουμε ποια είναι η πολιτική βούληση των δύο πλευρών για να δώσουμε ένα μήνυμα, να δώσουν ένα μήνυμα ότι θέλουν να ηγηθούν και να κινηθούν οι δύο πλευρές. Όπως σας είπα δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι η ώρα των αποφάσεων να δούμε κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση για να κινηθούμε. Σαν επόμενο βήμα, το... οι επεσταλμένοι του κουαρτέτου θα πάνε στην περιοχή, όλοι μας και οι τέσσερις. Εγώ ήδη βρίσκομαι εκεί, μένω εκεί με τον επεσταλμένο του ΟΗΕ και συνεργαζόμαστε επί τόπου, αλλά και με τις ΗΠΑ και με τους Ρώσους. Θα πραγματοποιήσουμε επισκέψεις, θα συνομιλήσουμε τις δύο πλευρές, να δούμε πώς μπορεί να προωθηθεί όλη η διαδικασία και αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Τρίτο, τελευταίο σημείο. Πώς να παραμείνει ανοιχτός ο πολιτικός ορίζον. Πολύ σημαντικό αυτό. Να βρούμε το σημείο εισόδου για την επανεκκίνηση αξιόπιστων διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα, αυτή η διαδικασία, η επιτόπια, ίσως είναι μια διέξοδος, είναι ένας τρόπος να πετύχουμε το στόχο μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα επιτόπου θα δημιουργήσουν μια όθηση, μια κίνηση. Να κινηθούν και οι ιδιωτέροι αλλά και οι άλλοι περιφερειακοί φορείς και εταίροι. Και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεω όσον αφορά το θέμα αυτό θα είναι σαφέστατη, διότι η θέση μας για τη λύση των δύο κρατών είναι σαφέστατη. Το γνωρίζετε όλοι. Νομίζω ότι τελευταίο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις ως αυτό σκοπό. Αυτό δεν θα ήταν κάτι χρήσιμο θα ήταν μάλιστα αντιπαραγωγικό. Χρειαζόμαστε σοβαρές προσπάθειες, επαφές, να προχωρήσουν τα πράγματα, ξεκινώντας από το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων να βελτιωθεί η κατάσταση του Παλαιστινίου σε επιτόπου και να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει. Εν κατακλείδη, αυτά είναι τα κεντρικά σημεία που ήθελα να παρουσιάσω. Βέβαια, με τα χαράς να συζητήσω μαζί σας και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις και εκεί θα έχω την ευκαιρία απαντήσεις να μπω σε λεπτομέρειες και πιο συγκεκριμένα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Τζετιλίνη για τις δράσεις του και για τα λόγια του σε ό,τι αφορά την ενευτική διαδικασία. Και εγώ συμμετείχα ε, συμμετέχω εδώ και τρία χρόνια περίπου σε αυτό το ζήτημα και έχω συναντήσει όλα τα ενδιαφέροντα μέρη και από την Ισραηλινή κυβέρνηση και από την Παλαιστινιακή Αρχή. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι επί της ουσίας οι λύσεις ε, γίνονται αποδεκτές ε, από τα δύο μέρη όταν μιλούμε ανεπισήμως. Είναι σχετικά κοντά και μάλλον διατεθειμένοι να κάνουν περισσότερες υπαναχωρήσεις από ό,τι παραδέχονται. Το πραγματικό πρόβλημα είναι το θέμα της εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν. Και από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και στις διαπραγματεύσεις αλλά και, στη... και ως εγγυητής γιατί πρέπει πραγματικά αυτά τα, αυτές οι εγγυήσεις να δοθούν ε, και από τις ε, δύο πλευρές. Και είναι περισσότερο ένας ε, συνασπισμός κρατών που θα κινηθεί προς αυτές τις εγγυήσεις και όχι τόσο ο ΙΕ και οι ανόκρανοι που θα είναι εγγυήτριες δυνάμεις, γιατί αυτό μου φαίνεται πραγματικό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή σας και να ακούσω και τη δική σας ανάλυση. Είναι το ζήτημα της ε, προβολής από τα μέσα. Εδώ και μερικά χρόνια, νομίζω 4-5, ήμασταν αρκετά κοντά. Ήδη υπήρχαν συνομιλίες με αμερικανική ε, διαμεσολάβηση και ένα από τα προβλήματα τότε ήταν ότι ο Αμερικανός εκπρόσωπος ενημέρωνε συνεχώς την τηλεόραση πιο συγκεκριμένα, ε, τα τηλεοπτικά μέσα για τις εσωτερικές συνομιλίες, κάτι το οποίο οδήγησε σε μεγάλες ε, αντιδράσεις ε, της κοινή γνώμης και οδηγηθήκαμε τελικά σε πάυση των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει εμπιστευτικότητα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχει γίνει πλέον κατανοητό αυτό από όλες τις πλευρές, αλλά και από ε, τους διαμεσολαβητές που αναφέρατε. Και κάτι άλλο το οποίο μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό ε, και δυσμενές είναι το παιχνίδι του τύπου και από την Ισραηλινή και από την Παλαιστινιακή πλευρά. που ε, διαδίδουν ακόμα και ψευδείς ε, ειδήσει, προσπαθώντας να προκαλέσουν την ένταση των συναισθημάτων και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόσκομα στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Αρχικά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τζεντιλίνη και να τον καλωσορίσουμε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θεωρούμε ότι είστε εταίρος. Ελπίζω και εσείς ε, να θεωρείτε ότι είμαστε εμείς εταίροι. Ξέρετε ότι είχαμε δύο συνομιλίες στην ε, Ολομέλεια ε, για την ειρηνευτική διαδικασία. Μάλιστα, στη μία από τι δύο ήταν και η κυρία Μογκερίνη. Επομένω, θα σα έχει ενημερώσει για τη γόνιμη αυτή συζήτηση που έγινε και ελπίζω να τα έχετε μελετήσει όλα τα όσα είπαμε εμείς εκεί. Σίγουρα το έχετε κάνει γιατί είστε γνωστός γι' αυτό. Υπήρξε ευρύτατη συνένεση στο Κοινοβούλιο, ελπίζω έτσι να σας βοηθούμε με το έργο σας. Πρέπει να υπάρχει ευρεία συνένεση σε ό,τι αφορά την ευτική διαδικασία στη Μεσανατολή. Γιατί αυτό είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε θετικοί απέναντι και στην κίνηση της κυρίας ε, Μογκερίνη, ε, διεύρυνση του κουαρτέτου, γιατί κάποιοι ε, θεωρούν ότι είναι αδρανές το κουαρτέτο και είναι θετική κίνηση να μπουν και άλλοι Άραβες εταίροι. Υπήρξαν πολλές αποτυχίες στο παρελθόν. Εύκολα μπορεί κάποιος να κολλήσει σε έναν κύκλο χαμηλών προσδοκιών. Όμως σε αυτή τη φάση η κυρία Μογκερίνη ε, έδειξε φιλοδοξία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας στηρίζει. Επομένως παρακαλούμε να διατηρήσετε το επίπεδο φιλοδοξιών παρό, παρόλα τα εμπόδια και τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε. Ξέρω ότι θα έρθουν και, και κατευθυντήρες γραμμές αυτή την εβδομάδα, ίσως και αύριο, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες. Ε, όχι ίσως γι' αυτό απλώς γιατί είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά για πλευρά πολιτικού αντικτύπου εάν αυτό θα επηρεάσει ε, και θα κινητοποιήσει περαιτέρω ε, την ειρηνευτική διαδικασία. Για την αύξηση της βίας. Προφανώς και η αποριστοκα... Ρίπο... <laughs> στην Ευρώπη ε, και μάλιστα μέσα Μέση Ανατολή είναι σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχετε κατά να μα πείτε σε ό,τι αφορά τι προβλέψει για την ειρηνευτική διαδικασία. Εμείς μιλούμε με την Παλαιστινική πλευρά και θέλουμε να υπάρξει αυτή η συμφιλίωση. Από την άλλη υπάρχουν σοβαρά εμπόδια ε, και από τους εκπροσώπους της ΦΑΤΑΧ και από το Εθνικό Συμβούλιο προκύπτει αυτό, όμως ε, και πάλι όσο μπορείτε εσείς να το αναδείξετε είναι σημαντικό. Ό,τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να σας στηρίξουμε θα το πράξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλίνη. Τρία σημεία μόνο συγκρατώ από την σύντομη παρέμβασή σας. Αν κατάλαβα καλά μιλήσατε για μια διαδικασία μεταμόρφωσης ε, για να ξαναπούμε στην πολιτική διαδικασία. Μίλησατε για τη Γάζα. Τι ακριβώς εσείς εννοείτε όμως. Μιλήσατε επίσης για ηγεσία. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια και για την Παλαιστινιακή ηγεσία. Γιατί ο Μαχμούτα Αμπάς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω μάλλον από τα μέσα, είναι μάλλον κουρασμένος. Ε, ε και κάποια στιγμή θα σταματήσει και αυτή η δράση. Επομένως, ε, τι λέτε, και, εφόσον μιλούμε δηλαδή για την ηγεσία, υπάρχει και η Παλαιστινιακή ηγεσία. Και δεν μιλώ για το πολιτικό στοιχείο εδώ και φτάνω έτσι στο τελευταίο. Δυστυχώς ε, το είδαμε αυτό ήταν μεγάλη ντροπή γιατί στην ολοπέλειά μας είχαμε η, λύση των δύο κρατών δεν ήταν η λύση των δύο κρατών για δύο λαούς. Ο, ο είχε δώσει αυτό και στον, ε, ε, στον τύπο. Είπε ότι δεν θα αναγνωρίσω ποτέ ένα εβραϊκό κράτος. Επομένως, για τον ίδιο θέλει να έχει Παλαιστινιακό κράτος για τον Παλαιστινικό λαό, αλλά όχι Εβραϊκό κράτος για τον Εβραϊκό λαό. Επομένω, δεν θέλει και πολύ μυαλό για να σκεφτεί κανείς ότι δεν πιστεύει σε αυτή τη λύση πραγματικά. Θέλει να είναι μόνο αυτό το αφεντικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με αυτή την προσέγγιση. Ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να σας πω όμως, δυστυχώς πέθανε σήμερα ο Χέλμουτ Σμιτ. Προερχόταν βέβαια από ένα πολιτικό κόμμα το εναντίον του οποίου είχαμε αγωνιστεί όλοι, αλλά ήταν ένας σημαίνων πολιτικός, έχουμε πολλά για τα οποία να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ο Χέλμουτ Σμιτ ήταν αποφασιστικός για να υπάρξει η άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλα αυτά τα οποία έγιναν με τη δυτή απόφαση του, του ΝΑΤΟ και με την εφεύρεση του νομισματικού φιδιού του πρόδρομου του ευρώ είναι στοιχεία τα οποία ανατρέχουν στις προσπάθειες του Χέρμου Σμιτ. Η κυρία Σακορά θα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλίνη, η Δυτική Όχθη, η Γάζα, η Ιερουσαλήμ έχουν μετραπεί σε πεδίο μάχη. Η Παλαιστίνη πρέπει να το παραδεχθούμε εξεγείρεται και εξεγείρεται με έναν μοναδικό τρόπο και για πρώτη φορά στα χρονικά τη ιστορία τη. τη δική, έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμή 72 Παλαιστίνοι πολίτε, 2.130 τραυματίστηκαν και 1.350 μπήκαν στη φυλακή. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό δεν θα σταματήσει αν δεν θα σταματήσει η μήτρα του κακού που είναι η κατοχή η καταπίεση, ο ρατσισμός, το apartheid, ο στραγγαλισμός των ελευθεριών και των δικαιωμάτων σε βάρος τους. Κύριε Τζελίδη Ντιλίνη, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει με τον τραγικότερο τρόπο την παταγώδη αποτυχία και το αδιέξοδο της ευρωπαϊκής πολιτικής για ειρήνευση στην περιοχή. Η απάντηση τη Επιτροπή και του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η πολιτική δέσμευση και η συμμετοχή είναι ο πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να μεταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ανησυχίες τη, στι αρμόδιες πλευρέ τη περιοχή, είναι προκλητική όταν το Ισραήλ έχει εμπράκτως αποδείξει ότι δεν θέλει καμία λύση. Έχουμε ακούσει όλοι, φαντάζομαι και εσεί, τον κύριο Νετανιάχου να αμφισβητεί τη λύση των δύο κρατών. Κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο, τη στιγμή που βλέπουμε τα παλαιστινιακά εδάφη, και αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε κύριοι συνάδελφοι όλοι εδώ μέσα, ότι εξαφανίζονται μέρα με τη μέρα και δορίζονται στους Ισραηλινούς επίκους. Για να φτάσουμε σήμερα, μετά τις αλλεπάλληλες μαζικές εκαθαρίσεις, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να συζητάμε για δεύτερη φορά την απαγόρευση της εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ισραηλινών προϊόντων που προέρχονται από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ε, λοιπόν, καλά κάνει ο κύριο Νετανιάχου και εγκαθίδει σε επιστολή του τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφαση αυτή, λέγοντα ότι τα γεωγραφικά όρια που εγγράφονται σε αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ είναι προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλόμενων μερών και ότι αν εφαρμοστούν θα πληγούν οι ευρωισραηλινέ σχέσει. Κύριε Τζεντιλίνη, εγώ θα καλωσορίσω την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων που έρχονται με καθυστέρηση αρκετών ετών, θα έλεγα, και περιμένω από το Συμβούλιο αλλά και από την Επιτροπή να προχωρήσουν στην εφαρμογή του άρθρου 79 της Σύνδεσης μεταξύ των δύο μερών και να καταγγείλουν αλλά και να την παγώσουν. Σας ευχαριστώ. Schmidt. Schmidt. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ε, δεν πρόσεξα. Κύριε Τζεντιλίνη, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, σας θεωρούμε βασικό συνομιλητή σε αυτές τις ε, συζητήσεις, αλλά βέβαια δύσκολα μπορεί κάποιος να ξέρει από, πού να ξεκινήσει κανείς. Και δυστυχώς έχασα και ένα τμήμα της ε, παρέμβασής σας, αλλά με ενημέρωσαν το περιεχόμενό της. Υπάρχουν τόσε εξελίξει αυτή τη στιγμή που δύσκολα μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει την ουσία. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι και οι δύο πλευρέ, και η Παλαιστινιακή Αρχή αλλά και η Ισραηλινή κυβέρνηση, ε, χάνουν ε, τον έλεγχο πολλών φορέων επιτόπου. Υπάρχει μια έλλειψη σεβασμού και αξιοπιστία ε, τη Παλαιστινική Αρχή στον Παλαιστινιακό λαό και από την άλλη και στο Ισραήλ ισχύει το ίδιο. Το 1993 είχαμε 2.000 ε, δυνάμει ε, εγκατάσταση των settlers. Ε, τώρα είναι 6.000 και εγώ ήμουν στην περιοχή πριν από. Ε, υπάρχουν 600.000 μάλλον. Και εγώ ήμουν στην περιοχή πριν από μικρό χρονικό διάστημα και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Και έτσι τα πράγματα δυσχεραίνονται, δεν διευκολύνονται. Ο κύριο Χάουιτ ανέφερε την παστιλινική συμφιλίωση τι είδου συζητήσει είχατε εσεί για να διευκολύνετε αυτή τη διαδικασία συμφιλίωση, Γιατί η ελλείψη αυτή τη συμφιλίωση, ε, η αξιοπιστία δεν υπάρχει. Αντίστοιχα, ε, και σε ό,τι αφορά την ε, αραβική-ισραηλινή κοινότητα, τι είδου συναντήσει είχατε με μέλη τη Κνέσετ και αν δεν έχετε κάνει τέτοιε συναντήσει, θα τι κάνετε γιατί είναι πολύ σημαντικοί και αυτοί οι συνομιλητέ. Ε, θα δούμε και τις καθηγητήρες γραμμές για την σήμανση ε, των ε, γεωργικών προϊόντων. Είναι υποκατοχή αυτά τα εδάφη, επομένως είναι παράνομα αυτά τα προϊόντα και στην αντίστοιχη περίπτωση της Κρυμαίας σταμάτησε η εισαγωγή των προϊόντων αυτών απευθεία και υπάρχουν κυρώσει. Και τώρα εδώ πέρα μιλούμε για κατευθυντήρες γραμμές μετά από τόσα χρόνια κατοχής. Βεβαίως τις περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το κατά πόσο θα επεκταθούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και ε, για να καλύψουν και άλλους φορείς ε, ή θα αφορά μόνο τα γεωργικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Thank you. Κύριος Κρυστάλτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Τζεντιλίνη για την παρουσία του εδώ σήμερα, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, ούτω ώστε να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να του θέσω τρει ερωτήσει πιο συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή σα, είναι δυνατόν να ξεκινήσει αυτή η πολιτική διαδικασία για αξιοπιστή διαπραγματεύσει που αναφέρατε με την παρούσα ηγεσία, βλέποντα ότι διάφορα μηνύματα και δείκτε μα κάνουν να πιστεύουμε ότι και οι δύο ηγέτε, οι παρόντε, είναι εν μέρει όμοιροι των ακραίων πτερίγων, πολλωμένων πτερίγων των ε, κομμάτων τους, δυνάμεών τους. Δεύτερο ερώτημα αφορά τον ρόλο των χωρών του κόλπου. Αναφερθήκατε σε μια συνεισφορά που θα μπορούσε να είναι θετική. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας σχετικά με αυτά που βλέπω διαβάζοντας και τα διεθνή άρθρα τα τελευταία χρόνια, τη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Μια συνεργασία πάρα πολύ στενή, αν τη δει κανεί από την πλευρά τη προσέγγιση όσον αφορά τη Συρία, αλλά κυρίω πιο γενικά την αντίθεση με τον υπαριθμό ένα εχθρό και τον δύο που είναι το Ιράν. Και έναντι των φιλοδοξιών των περιφερειακών τη χώρα αυτή και των πυρηνικών φιλοδοξιών. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, τι λέτε για τις δηλώσεις ε, κάποιων διπλωματών όπως του κυρίου Μάικλ Λόρεν που είναι ο πρέσβης του Ισραήλ στη ΣΥΠΑ ε, για το τι παίζεται στα παρασκήνια. Το παιχνίδι παίζεται στα παρασκήνια. Μήπως κατά κάποιο τρόπο μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ε, παρεμπόδιση επανέλεξη των διαπραγματεύσεων διότι η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να βασιστεί στην, ε, όταν βασίζεται στο Ισραήλ, ίσως να μην θέλει να συμβάλλει τόσο πολύ στην επανεκκίνηση της προσπάθειας εξέρευσης λύσης. Τελευταίο ερώτημα που αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η υποψή σα όσον αφορά την πιθανή αποστολή που θα μπορούσαμε να στείλουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, peacekeeping, ε, ειρηνευτική δηλαδή, στι ε, κατεχόμενες περιοχές και πιο συγκεκριμένα και στην Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, για να διατηρηθεί η ειρήνη και να αποφύγουμε και άλλες ε, βιοπραγίες. Είναι εφικτή αυτή η λύση. Τι συμβουλές συγκεκριμένες θα μπορούσατε να μας δώσετε επί του συγκεκριμένου. Ευχαριστώ. Σφάιφερ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Σλάιφερ από την Ολλανδική Γερουσία. Θα μιλήσω τη μητρική μου, αν σα πειράζει. Θα ήθελα λοιπόν ε, να θίξω το ζήτημα τη ελευθερικής Διαδικασία ε, στη Μέση Ανατολή. όπω ανέφερε ο κύριο Τσιντιλίνη, είναι πιο επίγον από ποτέ αυτό το ζήτημα, υπό το φως και της πολιτικής αστάθειας ε, στην ευρύτερη περιοχή. Το ερώτημα μου είναι αν ο ειδικό εκπρόσωπος έχει την γνώμη ότι εξακολουθεί να είναι η καλύτερη λύση η λύση των δύο κρατών τώρα που αυτή η ιδέα του ενός ε, διεθνοτικού ε, κράτους, παρότι για το Ισραήλ έχει πρακτικές ε, προεκτάσεις και προβλήματα, γι' αυτό και δεν θεωρείται ρεαλιστική. Εγώ έρχομαι από τη Χάγη και πολλές φορές εξετάζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η γενική σύγκρουση να ελεγχθεί και από βάση νομικού πλαισίου και έτσι να βρούμε μια ειρηνευτική διαδικασία και λύση. Έχουμε τέσσερι ακρογωνιαίου λήθους. Πρώτον, το κείμενο δίκαιο του κράτους τη Ισραήλ. Δεύτερον, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του Παλαιστινιακού λαού. Τρίτον, τα δικαιώματα και υποχρεώσει των δυνάμεων κατοχής. Και τέταρτον, οι κανόνε ε, σε ό,τι αφορά την χρήση βία, συμπεριλαμβανομένη και τη αρχή τη αναλογικότητα. Τώρα, Πρόεδρε, ε, αυτό το νομικό πλαίσιο περιγράφεται λεπτομερώς ε, στο Advisory Opinion, στη συμβουλευτική νομοδότηση του Διεθνούς ε, Δικαστηρίου θεωρείται του τείχους του Ισραήλ. τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί το πρόσχημα ή τουλάχιστον διατείνεται ότι ακολουθεί το soft power και τώρα που έχει σταματήσει η Αμερικανική ε, ειρηνευτική πρωτοβουλία ή τουλάχιστον δεν έχει αποτελέσματα, τότε ποια θα είναι η ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως πρέπει να κάνει περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της ως ε, δύναμη διευκόλυνσης ή διαμεσολάβησης στην ειρηνευτική διαδικασία. Ποια είναι η δική σας γνώμη γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία έχει ως σκοπό την ε, προετοιμασία ε, μιας ε, καλής διαδικασίας για να συμφωνήσουμε επί των παραμέτρων και των τελικών όρων μιας ειρηνευτικής συμφωνίας εντός αυτού του νομικού πλαισίου του Διεθνούς Δικαστηρίου. Πώς θα διατυπωθεί αυτό και πώς θα καταλήξουμε στη τελική συμφωνία. Αυτό είναι το κύριο ερώτημά μου προ ε, τον ειδικό εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Ειδικό εντεταλμένο, συγγνώμη. Κύριε Βανόρντεν. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε για μια ακόμα φορά από αυτά που είπε ο κύριος Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον υποστηρίζει, είπε, μια λύση δύο κρατών. Είπε ότι, ότι θέλει να έχει ένα Ισραήλ και ένα αποστατικοποιημένο Παλαιστινιακό κράτος το οποίο αναγνωρίζει το Ισραηλινό κράτος. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Παλαιστινιακής Αρχής, είσαστε ικανοποιημένος ότι ασκούμε την πρέπουσα πίεση σε αυτούς τους Παλαιστίνιους για να τους πείσουμε να επανέλθουν στη διαπραγματευτική τράπεζα. Οι Ζαρινοί με τον Νετανιάχου είπαν ότι είναι έτοιμοι να περάσουν σε διαπραγματεύσεις και με χωρίς όρους κιόλας. Είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις αυτοί που δεν θέλουν να διαπραγματευτούν είναι οι Παλαιστίνοι. Τι θα κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Ο κ. Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχουν πολλοί σε αυτή την αίθουσα συμπεριλαμβανομένου και του κ. Τζατιλένη ότι πραγματικά το Ισραήλ ενδιαφέρεται να βρεθεί λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα εάν αυτή είναι η εντύπωση σε οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Πλανάτε πλάνην μεγάλη. Ο μόνος τρόπος, αν θέλουμε να δούμε πιθανή διέξοδο, είναι οι κυρώσει εναντίον του Ισραήλ. Πράγμα το οποίο δεν συζητά κανένα. Κανένα από όσου έχουν τη δυνατότητα να το, να το κάνουν. Το Ιράν, για παράδειγμα, ήρθε σε κάποια διαπραγμάτευση με τη διεθνή κοινότητα γιατί μπήκαν κυρώσει. Πώς αναμένουμε το Ισραήλ να συζητήσει στα σοβαρά με τη διεθνή κοινότητα την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος, εάν δεν σκεφτούμε τρόπους που να αναγκάσουν το Ισραήλ να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω κάτι λέει ένας συνάδελφος, αλλά δεν ξέρω τι λέει. Ε, καταλήγω λοιπόν ότι εάν θέλουμε πράγματι να δούμε πιθανή διέξοδο σε αυτό το ζήτημα, είναι να είμαστε σοβαροί ας πούμε το Ισραήλ δεν έχει πυρηνικά όπλα. Γιατί δεν γίνεται συζήτηση για αυτό το πράγμα. Είναι, είναι όποιος προλάβει πρόλαβε. Γιατί έτσι φαίνεται είναι. Όποιος προλάβει πρόλαβε. Έχω κλείσει αυτή ήταν η παρέμβασή μου. Θέλω να δω από τον εκπρόσωπο εδώ της, ε, της Κομισιόν αν υπάρχει πουθενά οποιαδήποτε συζήτηση να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τσεντιλίνη, εγώ ενοχλούμε από την αύξηση της βίας και οι επιθέσεις στους Ισραηλινούς δρόμους που έχουν γίνει πρόσφατα πρέπει να καταδικαστούν από όλους. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι το Ισραήλ ήταν υποχρεωμένο να κάνει να οδηγήσει σε περιορισμού, να οδηγηθεί σε περιορισμού και ζητούμε από τους Παλαιστίνους να σταματήσουν την εχθρική ρητορική του. Πρέπει το Ισραήλ να έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Δεν χρειάζεται πια να, είμαστε, να δεχόμαστε τους απολογητές της Χαμάς. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για διάθεση της Χαμάς να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ινδία είπε μήπως πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα της ύπαρξής τους. Αλλά και δεν υπάρχει κάποιος Παλαιστινίος που να μην δέχεται το δικαίωμα της, την ύπαρξη του Ισραήλ, επομένως και το δικαίωμά του να υπάρχει. Αλλά για τους Παλαιστινίους αυτό δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται. Δεν δείχνει λοιπόν το πραγματικό δίλημα. Εμείς ε, εξακολουθούμε να ε, επικρίνουμε το Ισραήλ τη στιγμή που δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμα το δικαίωμά του να υπάρχει. Για να έχουμε πρόοδο, λοιπόν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την αναγνώριση του δικαίωματος του Ισραήλ να υπάρχει. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Τζεντιλίνη. Και εγώ πιστεύω ότι η λύση δύο κρατών είναι σημαντικό και κέριο στοιχείο στι διαπραγματεύσει. Δεν υπάρχει λύση στην περιοχή αυτή χωρίς μια επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών, αποδεκτής ε, λύσης. Το ερώτημα μου όμως είναι το εξή. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβει τετραμερή στο μέρο το κουαρτέτο. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει το κουαρτέτο να έρθει σε επαφή και με τους Ισραηλούς και τους Παλαιστινίους στις επόμενες εβδομάδες. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την διεθνή αντιμετώπιση της κρίσης. Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ισραήλ. Κατά την βάση της δικής σας εμπειρία θα ανταποκριθεί σε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωση στο Ισραήλ και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε καλύτερη συνεργασία του κουαρτέτου με, την, με τον Αραβικό Σύνδεσμο και αν ο Αραβικός Σύνδεσμος θα είναι έτοιμος να απαλύνει τη μονομερή του θέση κατά του Ισραήλ. Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύετε ότι είναι κάτι περισσότερο από κενές υποσχέσεις. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ κύριε Σκάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλίνη, θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα εδώ σήμερα και την ε, παρέμβασή σα. Προφανώ πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα με πολύ μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο. Και ξέρετε, κάθε φορά που υπάρχει μια συζήτηση ακούγονται κάθε είδους επιχειρήματα από κάθε πλευρά. Όμως, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε το σύνολο της ε, κατάστασης, Ορισμένα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα ξεκάθαρα. Πρώτον, οι απώλειες αφορούν κυρίως την Παλαιστινιακή πλευρά. Βεβαίως υπάρχουν και απώλειες και από την Ισραηλινή πλευρά. Αλλά αν δείτε όλο το ιστορικό, είναι σαφές. Και το δεύτερο, αυτή η γη, αυτή η περιοχή, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαμάχη. Το Ισραήλ κατήχε 35% ε, των εδαφών και το υπόλοιπο 65% το είχαν οι Παλαιστίνοι. Και σήμερα, αν δείτε τι συμβαίνει στην πράξη, έχει αντιστραφεί η εικόνα. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει το 65% περίπου και η Παλαιστίνη περίπου 35%. Και με την διαστηριότητα των επίκων, τη συνεχή του διαστηριότητα, βλέπουμε ουσιαστικά ότι αυτή η ιδέα των, της λύσης των δύο κρατών πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας. Τελικά λοιπόν το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τους παράνομους επικισμούς που καταστρέφει στιγμή προς στιγμή την λύση των δύο κρατών και δεύτερον τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε ελπίδα και στην Παλαιστινική πλευρά. Γιατί αν δείτε πόσο έχουν υποφέρει εκείνοι, εκείνοι είναι ουσιαστικά που έχουν τραβήξει τα περισσότερα αν θέλετε. Και γι' αυτό με βάση και όλο το προσφυγικό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, πήγα εκεί πέρα σε προσφυγικό καταβλισμό και συνάντησα μια Παλαιστινική οικογένεια ε, όπου ήταν στον καταβλισμό τρεις γενιές. τρεις γενιές σε μία τέντα. Ένα νεογέννητο που γεννήθηκε στο Αρεμπίλ και η μητέρα του είχε γεννηθεί σε άλλο καταβλισμό στο Χαλίντ και η μητέρα της, η γιαγιά δηλαδή, είχε γεννηθεί σε άλλο καταβλισμό στη Βαλαιστίνη και μετά είχε μετατοπιστεί. Πρέπει λοιπόν, λοιπόν κάποια στιγμή να δώσουμε ελπίδα και στον Παλαιστινιακό λαό για να διατηρήσει αυτό το, κατάλογο που θε... το διάλογο που θέλουμε και να φτάσουμε τελικά σε μια λύση. Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν μπορείτε να απαντήσετε. Πότε θα έχουμε τις κατευθύνες γραμμές για την σήμανση ε, των προϊόντων που προέρχονται από τις ε, περιοχές αυτές. Ο κ. Παπαδάκης. Κύριε Τζεντιλίνη, ε, η τοποθέτησή σας ήταν στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιχείρηση, τη συστηματική επιχείρηση αποχαρακτηρισμού του ζητήματος, του προβλήματος του Παλαιστινιακού ακριβώς στην προσπάθειά σας να αποκρύψετε ότι υπάρχει κατοχή στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα και ακριβώς προσπαθώντας να αποχαρακτηρίσετε λοιπόν το πρόβλημα συνεχίζετε τη γνωστή τακτική Δηλαδή να θεωρείται ότι είναι ίσο, να εξισώνεται δηλαδή το θήτη με το θύμα. Όταν κατηγορείται για παράδειγμα ένας λαός που αγωνίζεται ενάντια στη βαρβαρότητα, ενάντια στο τείχος, ενάντια στους παράνομους επικισμούς, ενάντια στις ε, χιλιάδες φυλακής πολιτικών κρατουμένων ως τρομοκράτης. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν διαρκώς τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν με το κράτος του Ισραήλ και όταν έχει τεράστιες ευθύνες και η ελληνική κυβέρνηση που μόλις ολοκλήρωσε κοινή στρατιωτική άσκηση την Blue Flag με το Ισραήλ που επί της ουσίας αποτελεί προθέρμανση για νέες επιθέσεις σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Πώς τοποθετείστε απέναντι στο ζήτημα της κατοχής και στο ζήτημα της προκλητικής εξίσωσης του θήτη με το θύμα. Γιατί πρέπει να δοθεί λύση με ανεξάρτητο βιώσιμο ε, κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 67 δίπλα στο Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε εσά τα συμπεράσματα και τα καταστικά σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή συζήτηση, έτσι άκουσα τα επιχειρήματα όλων σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται σε περισσότερα από τα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρατε. Και όσο γίνεται πιο σύντομα να απαντήσω. Πρώτα να απαντήσω στην κυρία Λιο Μαγή, η οποία έχει φύγει το μεταξύ, αλλά νομίζω ότι έθιξε ζητήματα με τα οποία συμφωνώ πλήρως μίλησε για αποδεκτές λύσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η παρατήρηση, γιατί αν δείτε την ε, ευρύτερη περιοχή, ουσιαστικά υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις, τόσα εκρεμή ζητήματα. Αν δείτε αυτό το μέρος της περιφέρειας, της περιοχής, δηλαδή την ερευνητική διαδικασία Παλαιστίνης και Ισραήλ, υπάρχει η λύση. Είναι η λύση των δύο κρατών. Το αναφέρατε κι εσείς. Όλοι ξέρουμε προς τα πού θα πρέπει να κινηθούμε. Πράγματα λοιπόν δεν απέχουμε και πολύ, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο κύριος Χάουιτ είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Για τον αντίκτυπο του ε, τη ονομασία προέλευση, ε, που δεν είναι μποϊκοτάρισμα, απλώ ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και αυτό αφορά την ε, εφαρμογή τη ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν είναι τίποτα καινούριο. Υπάρχουν ήδη αυτοί οι κανόνε. Σημαντικό ήταν και το στοιχείο της συμφιλίωσης που ανέφερε και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα, παρότι υπάρχουν περιορισμοί και σε αυτό, γιατί υπάρχει βεβαίως η πολιτική και την τηρώ απολύτως την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συνομιλώ λοιπόν με τη Χαμάς. Βέβαια, το ζήτημα τη ε, συμφιλίωση είναι ένα θέμα το οποίο θίγω κάθε φορά ε, όταν πηγαίνω στη Ραμάλα, το θίγω ε, με την Παλαιστινική Αρχή όταν συνομιλώ. Μου λένε ότι το προάγουν γενικά, υπάρχει κάποια δέσμευση, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουν και άλλα πράγματα. για να ενισχύσουν την παρουσία τους ε, ε, στη Γάζα. Και ίσως αυτό να είναι και η αφετηρία της όλης διαδικασίας. Ο κύριος Μπέλντερ τώρα είπε κατά πόσο αυτοί είναι οι ηγέτες. Μήπως ε, παρατηρούνται στοιχεία κόπωσης. Το θέμα είναι ότι όλοι οι ηγέτες θα πρέπει να δείχνουν ηγετικό πνεύμα. Ποια είναι η λύση. Κάποιοι το αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σαφή ιδέα ε, περί τίνος πρόκειται. Μιλούμε για την λύση των δύο κρατών με τα σύνορα του 67. Εδώ βρισκόμαστε. Η κυρία Σακοράφα. Εγώ προσπάθησα να πω ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη βία που παρατηρείται στην περιοχή. Και επίσης ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε, ελέγχουμε την πολιτική βούληση να επιληθεί αυτή η κρίση με πολιτικά μέσα. Βλέπω και κατανοώ τα όσα βλέπετε κι εσείς. Αλλά αν θέλουμε να βοηθήσουμε, να έχουμε μια ωφέλιμη συμβολή, πρέπει να πιέσουμε οι ηγέτες να αξιοποιήσουν την ηγετική τους θέση και να κάνουν ένα θεραλέο βήμα προς τα μπρος. Το ανέφερα και πριν με βάση με τα όσα εμείς κάναμε για να προχωρήσουμε και ότι μπορούμε έτσι ε, με μια τέτοια συμφωνία να ε, ενισχύσουμε και τους ε, ε, Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Ο κύριος Σμιτ επίσης αναφέρθηκε στην ε, συμφιλίωση. Είναι σημαντικό και αυτό. Αυτή είναι η συνεχής μας προσπάθεια. Αναφερθήκατε και εσείς ε, στην ονομασία προέλευσης. Είναι κάτι το οποίο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και θα δούμε πώς αυτό το μέτρο θα επηρεάσει τα πράγματα. Τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα όσα μπορούμε να κάνουμε για να σημειώσουμε πρόοδο. Τα θα δούμε από εκεί πώς θα συνεχίσουμε. Ελπίζω να υπάρξει η πρόοδος. Ο κύριος Καστάλντο αναφέρθηκε το ρόλο της παρούσης ηγεσία και τις δυνατότητες που έχουμε. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες το να συνεργαστούμε και να εργαστούμε με αυτό που έχουμε στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από αυτό που διαθέτουμε. Ο ρόλος των χωρών του κόλπου, των περιφερειακών χωρών, των περιφερειακών εταίρων είναι σημαντικότατος. Και μεταξύ αυτών των χωρών σαφώς η Αίγυπτος έχει ρόλο όσον αφορά τη Γάζα, η Ορδανία όσον αφορά ε, άλλες περιοχές, η Σαουδική Αραβία έχει ρόλο να παίξει διότι κατά κάποιο τρόπο ήταν εκείνη που ξεκίνησε την ειρηνευτική ε, διαδικασία, την Arab Peace Initiative. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό της εντολής μου αυτή η ειρηνευτική διαδικασία και πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε είναι σημαντικό αυτή η αραβική πρωτοβουλία για την ειρήνη να είναι επιτάπητος. Νομίζω ότι είπα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι χρειάζεται να προωθήσουμε για την ώρα και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το κουαρτέτο και τους εταίρους της ε, αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουν. Νομίζω ο κ. Σρίβερ αναφέρθηκε σε κάτι που συμπεριλαμβανόταν ήδη στην απάντησή μου. Αυτή η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η δυνατή λύση. Και εμπολείς αυτό που βλέπετε εσείς επιτόπου, αυτή η βία εκεί επιτόπου, ίσως περαιτέρω δείχνει ότι πρέπει να πάμε προς τη λύση των δύο κρατών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ελέγχει αυτό το θέμα και έχουμε μέσα να υλοποιήσουμε αυτή την λύση επιτόπου. Ο κ. Βανόρντεν αναφέρθηκε σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό ο κύριος Νετανιάχου και αν χρησιμοποιούμε την πίεση που μπορούμε την επιρροή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε και με τι δύο πλευρέ. Αυτό είναι πολύ ξεκαθαρό. Αυτό που ζητούμε και από τι δύο πλευρέ, που και οι δύο θέλουν τις δύο, τα δύο κράτη, είναι να το μεταμορφώσουν αυτό στην πράξη. Και έχουμε όλα τα μέσα για να το στηρίξουμε αυτό, αν το αποφασίσουν εκείνοι να κινηθούν προς τα εκεί. Νομίζω ότι έχουμε μια φωνή, έχουμε ένα ρόλο Νομίζω ότι υπάρχει πολιτικό περιθώριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Χατζηγεωργίου ρώτησε κατά πόσο ενδιαφέρεται στην ειρήνη, για την ειρήνη του Ισραήλ και αυτό το σχόλιο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να πιέσουμε να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία. Διότι αυτή η διαδικασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και ο κύριος Κάμπερ ε, διερωτήθηκε κατά πόσο το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Εγώ παραπέμπω στην Αραβική Πρωτοβουλία για την Ειρήνη. Αυτό είναι σημαντικό που έχουμε. Αυτή η πρωτοβουλία εμπεριέχει πολλά εκφράζει το περιφερειακό συνέστημα. Υπάρχει προσφορά, επιτάπητος, νομίζω ότι είναι σημαντική βάση για μας για να σημειώσουμε κάποια πρόοδο μέσω διαδικασίας. Ο κύριος Πώς ρώτησε ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα. Προσπάθησα να τα αναφέρω, δεν θα ήταν χρήσιμο να παραθέσω κατάλογο πραγμάτων που ήδη υπάρχουν, είναι γραμμένα εμπεριέχονται στη δικασία του Όσλο σαν παραρτήματα. Αυτό που εξετάζουμε είναι να δώσουμε δύναμη, μεγαλύτερη δύναμη στους Παλαιστινίους στη Δυτική ε, Όχθη και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Ισραήλ μέσω υποδομών, οικονομικής ενισχύσεως, βοήθειας για την ενίσχυση ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις ανάγκες των δύο πλευρών. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία, αν επιτευχθεί πρόοδος, τότε μπορούμε να βρούμε περισσότερα πράγματα. Η όλη περιοχή μπορεί να βρει περισσότερες λύσεις. Και αναφέρθηκα στην αραβική ειρηνευτική διαδικασία, ο κύριος στην ιστορία. Ε, εγώ τίνω να βλέπω σε τι μπορώ να είμαι χρήσιμος εκεί, επί τόπου. Θέλω να βοηθήσω. Αυτή είναι η μόνη μου μικρή φιλοδοξία. Θέλω να βοηθήσω. Η ιστορία κατά την άποψή μου δεν βοηθά νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Ε, η διάταξη που αναφέρατε, η διατάξη που αναφέρατε και οι προβλέψεις έχουν δρομολογηθεί. Νομίζω, α, στον κύριο Παπαδάκη να απαντήσω. Ξανά θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια θέση. Είναι σαφές. Αναφερθήκατε σε αυτή. Δύο κράτη είναι η λύση να επανέλθουμε στα σύνορα του 67. Αυτό που είπατε. Δεν θέλω να κρύψω τίποτα. Νομίζω ότι έχω πολλά να πω εκεί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να πει πάνω σε αυτά. Λίγο πολύ εδώ βρισκόμαστε και ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Ζεντιλίνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να ξαναμιλήσουμε. Δυστυχώς το θέμα αυτό δεν λύνεται τώρα εδώ. Ευχαριστώ πραγματικά που ήρθατε. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Στο επόμενο σημείο που έχουμε. Α, ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό. Uh, the passing uh, away of major statesman Απεβίωσε ένας μεγάλος ηγέτης, ο Χέλμουτ Σμιτ, uh, όπως είπατε, ήταν πολύ σημαντικός για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Εξελίξεων. Ίσως θα έπρεπε να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ε, προς τιμήν και εις μνήμη του καγκελαρίου Σμιτ που ήταν τόσο σημαντικός άνθρωπος. Εγώ προέρχομαι από το ελληνικό κοινοβούλιο, δεν ξέρω ποιο είναι το πρωτόκολλο εδώ. Εγώ θα θεωρούσα ότι είναι σημαντικό να ε, τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα τόσο μεγάλο ηγέτη. The session Uh, e Κοιτάξτε, μιλήσαμε τώρα για τους πολέμους αντιπροσώπων στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ε, θα καλέσω τον, είχα καλέσει τον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, τον καλωσορίζω αυτόν και του συναδέλφους του που ήρθαν και θα ακολουθήσω τη συμβουλή του Έλληνα συναδέλφου μας, δηλαδή θα ήθελα να ζητήσω από σας να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή, να προσευχηθούμε και να σκεφτούμε τον Helmut Schmidt, προς τιμή του Helmut Σμιτ. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Ε, λοιπόν, σχετικά με τους πολέμους διαντιπροσώπων στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημόσια κρόση και ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το κάναμε ήδη στην προσέγγισή μας όταν συζητήσαμε το θέμα με τους συναδέλφους των Βαλκανικών κρατών. Ε, και έχουμε επιστήμονες για να συνεχίσουμε, κυρίως για τα θέματα που άπτονται της Μέσης Ανατολής. Ακούσατε τη θέση μου σήμερα το πρωί. Δεν θα επαναλάβω αυτά που σας είπα και θα ήθελα να δώσω αρκετό χρόνο στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Στρέφοντας γύρω μου, δεν βλέπω να είναι εδώ όλοι οι ομιλητές. Ο κ. Βόλτσουκ, η κυρία Βόλτσουκ μάλλον. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι πρώτος? Δόκτωρ Καμί Πεκαστάν είναι ο πρώτος στους ομιλητές. Είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα, πρόγραμμα για τη Μέση Ανατολή στο, στο σχολείο John Hopkins στην Ουάσιγκτον και θα ήθελα να ζητήσω να ξεκινήσει με δηλώσεις με αυτά που έχει να πει. Έχει στη διάθεση του ένα δεκάλεπτο περίπου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκτός μικροφώνου. <clears throat> Το πρώτο θέμα είναι ο ίδιο ο πόλεμος αντιπροσώπων, δεν υπάρχει κάτι καινούριο εδώ. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από τότε που υπάρχει πόλεμος. Ωστόσο, ένα παράδειγμα και στην Αμερικανική Επανάσταση ξεκίνησε ως πόλεμος αντιπροσώπων ε, μεταξύ Γάλλων και Άγγλων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του, Α, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη, λέει ο κύριο Μπροκ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Είναι αυτό το φίλτρο αποφεύγουμε ουσιαστικά την κλιμάκωση. Ένα καλό παράδειγμα ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Είχαμε πόλεμους για προσώπων στον ψυχρό πόλεμο, γιατί, στο ψυχρό πόλεμο, γιατί δεν ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις να υπάρξει πραγματική μετοπική επίθεση εξαιτία ε, της πυρηνικής απειλής. Γι' αυτό είχαμε δεκάδες ε, τέτοιους ε, πολέμους μετά το 1945. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ο έλεγχος του κόστους γιατί έχουμε σύγκρουση χαμηλής έντασης, όπου η μεγάλη δύναμη χρησιμοποιεί έναν ε, αντιπρόσωπο μικρότερου μεγέθους, ε, με χαμηλότερο κόστος, πολύ περιορισμένο κόστος, σε μια επικράτεια που μπορεί να υπάρχουν πόροι, υπάρχει δίωδος ε, εισόδου και μπορούν έτσι να το ελέγξουν περισσότερο. Το, δε, το τρίτο πλονέκτημα είναι αυτό που αποκαλώ η παγίδα ένας ασύμετρος πόλεμος για προσώπων. Εδώ εννοούμε το ασύμετρο κόστος ε, των κανονικών έναντι των μη κανονικών δυνάμεων. Η αναλογία μπορεί να είναι 1 προς 100 ή ακόμα και 1 προς 1000 ή ακόμα παραπάνω. Αυτό επιτρέπει ε, να απομυζήσουμε οικονομικά τον, ε, τον αντίπαλο. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, η Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν 1980, άλλα παραδείγματα μεταξύ του 2003 και 2012-2013, ε, στους πολέμους Αφγανιστάν και Ιράκ. Το κλειδί εδώ, σε αυτή την παγίδα, είναι να ε, παγιδεύσουμε τον αντίπαλο, δηλαδή να τον ε, προσελκύσουμε να δίνει τακτικά δυνάμεις ε, και έτσι τον αποδυναμώνουμε οικονομικά. Τώρα, για το... Ναι. Μιλούμε περισσότερο για την περιφέρεια και όχι τόσο για συγκεκριμένα κράτη. Θα μιλήσω μόνο για τους ε, περιφερειακούς ε, ε, φορείς και όχι τόσο για τους αντιπροσώπους, ούτε για τις μεγάλες δυνάμεις. Θα αναφερθώ στη συνέχεια. Για το Λεβάντε μιλάει ο μιλητής συγκεκριμένα. Ε, έχουμε διάφορες δυνάμεις, Ισραήλ, η Ιορδανία, είναι ε, ιδιαίτερα επιφυλακτικέ, δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα, κοιτάζουν από, ε, από το πλάι, όμως πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Πιο ενεργοί φορεί τώρα είναι η Τουρκία που πάντα έτσι, έχει μια πολύ στεναρή παρουσία, εμπλέκεται και στην προσφυγική κρίση και στη στήριξη των αντιπροσώπων στη Συρία, όμως η ίδια Τουρκία δεν έχει μεγάλη ισχύ περιφερειακά πιο πολύ ε, εμπλέκονται η Σαουδική Αραβία και τα Αραβικά, ε, Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ. Όμως δεν εμπλέκουν ε, τακτικές δυνάμεις. Η μη περιφερειακή δύναμη που πραγματικά εμπλέκεται είναι το Ιράν και ο περιφερειακό δορυφόρος που είναι η Χεσβολάχ. Το Ιράν έχει μακροπρόθεσμη ε, συμμαχία και με την Χεσμολά από την δεκαετία του 80 και αυτό δεν έχει αλλάξει από τότε και έχει ε, οδηγήσει το Ιράν στο να εμπλέκει τακτικές δυνάμεις στη Συρία. Αυτή η δέσμευση επιτρέπει στη Σαδική Αραβία και στους, στις δορυφορικές δυνάμεις ε, να κάνουν αυτόν τον πόλεμο για την προσώπων και έτσι απομιζούν οικονομικά τους Ιρανούς ε, στη σύγκρουση στη Συρία. Όμως ε, ήταν πιο έξυπνο το Ιράν ε, σε αυτό που έγινε στην Ιεμένη και βλέπετε ότι οι Ιρανοί ασχολούνται με τη Συρία ενώ οι Σαουδάραβες στην Ιεμένη. Και έτσι έχουμε όλο αυτό το απομακρυσμένο παιχνίδι, όπου ο ένας ασκεί πίεση στον άλλον και ουσιαστικά οδηγεί ο ένας τον άλλον στη χειροκοπία περιφερειακά. Αυτή η διαμάχη όμω γίνεται σε ένα πλαίσιο όπου οι τιμέ του πετρελαίου είναι πολύ χαμηλέ και έτσι και οι δύο οικονομίε είναι πολύ αδύναμε και έχουν πολύ μεγάλο εσωτερικό πολιτικό ρίσκο. Και είναι δύσκολο να κάνει κάποιο πόλεμο πέρα από τα σύνορά του όταν έχει πολύ χαμηλά έσοδα. Αυτή η διαμάχη εξηγεί και τι ε, συγκρούσει μεταξύ Σαουδική Αραβία και Αμερικανών εταίρων γιατί η πυρηνική συμφωνία που έκανε οι Αμερικανοί με το Ιράν ε, δίνουν πόρους στο Ιράν που αλλιώς δεν θα ήταν διαθέσιμοι και διευκολύνει και την θέση ε, των ΗΠΑ απέναντι στην Σαουδική Αραβία. Και έτσι φτάνω στις ΗΠΑ και στην πολιτική τους ε, απέναντι στο Λεβάντε. Ε, πρώτον, βρισκόμαστε εν εκλογών του χρόνου, επομένω δεν ασχολείται κανένα με την εξωτερική πολιτική. Πολλοί όμως επικρίνουν ότι η πολιτική είναι αντιφατική, αναποτελεσματική, κατακρίνουν κυρίως ε, τον Ομπάμα και τη Σούζαν Ράι. Ο ίδιο ο πρόεδρο. Ε, ασχολείται με την εξωτερική πολιτική κυρίως ό,τι αφορά το κληροδότημά του. Αρχικά έχει την πολιτική του να μην κάνει τίποτα χαζό. Μετά ήθελε να επικεντρωθεί ε, στα, στα όπλα μαζικής καταστροφής στην περιφέρεια και η κύρια πολιτική του ήταν να κάνει ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τρομοκρατική επίθεση είτε σε αμερικανικό έδαφος ή κατά των αμερικανικών συμφερόντων. Η τρίτη τρομοκρατική απειλή οδήγησε την αμερικανική πλευρά να επικεντρωθεί στον ISIS και έτσι έχει, αυτή, ε, αναπτύξει αυτή την αιμονή με τον ISIS που έχει λειτουργήσει υπέρ του Ιράν και ε, αυτού του καθεστώτος. καθώς ε, και ε, αξιοποιήθηκε αυτό το στοιχείο της συμφωνίας με όπλα από το Ιρανικό και από το Συριακό καθεστώς. το άλλο στοιχείο που ανέφερα, το να μην κάνει κάτι χαζό σε ανόητες επιθέσεις, μάλλον κινήσεις, έχει οδηγήσει σε μία ε, λιπόψυχη, αν θέλετε, προσέγγιση οι ΙΠΑ έχουν υπονομεύσει τη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι σε σημείο ρήξη. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι ουσιαστικά. Ε, το, έχει αλλάξει την πολιτική το απέναντι στο Ιράν, αλλά δεν ε, είναι και εταίρο ακριβώς. Επομένω, είναι μια τέτοια μεσοβέζικη κίνηση που έχει ακολουθήσει. Καμία χώρα τη ευρύτερη περιοχή δεν είναι πραγματικά εταίρο εμπιστοσύνη, ούτε και αντίπαλο οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αντιπροσώπους ε, στη Συρία μέσω του προγράμματος Train and Equip, κατάρτισης δηλαδή, όμως με πολύ περιορισμένο ορίζοντα και δεν έχουν δυνατόν να κάνουν τίποτα που να οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων. απλώ περιορίζουμε κάπω ε, τις ζημίες ε, χωρίς προοπτική για το μέλλον. Και για να φτάσω στο τελευταίο μου στοιχείο είναι οι συστάσει πολιτική πολιτική για οικονομική περιορισμοί για κάθε μεγάλη δύναμη είναι τεράστια και για την ΣΥΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγα χρόνια μετά την οικονομική χρηματοστατική κρίση μάλλον δεν υπάρχει όρεξη, διάθεση να κάνουμε πολλά για να αλλάξουμε την πορεία της περιοχής. Ακόμα και αν υπήρχε βούληση δεν υπάρχει καλή πολιτική. Υπάρχουν μόνο τεράστια ρίσκα με, με πολύ μεγάλο κίνδυνο ζημίας. Και το επόμενο στοιχείο είναι ότι ακόμα και αν υπήρχε πολιτική, είναι αδύνατον κάποιο να ελέγξει το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει, είναι ιδιαίτερα ασταθή η περιοχή και δεν υπάρχουν καθόλου εγγυήσει. Πρέπει κάποιο να είναι πολύ ευέλικτο για να προσαρμόζεται τις εξελίξει της περιοχής. Τελευταία στοιχεία για τη σύσταση. Ε, να κινηθούμε με ένα πολύ ανοιχτό και ευέλικτο πνεύμα. Ουσιαστικά έχουμε ε, τα 100 χρόνια μετά την ίδρυση του Λεβάντα, ίσως θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την αναφορά και να εξετάσουμε με ανοιχτό πνεύμα την πολιτική δομή εκεί της ε, Ανατολής. Τα πράγματα θα αλλάξουν αν το Ισραήλ και η Ορδανία αλλάξουν στάση και αν ε, μπουν σε δυσκολίε, ε, τότε θα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε πραγματικά ανακατανομή και ανασχεδιασμό τη ευρύτερη περιοχή που να επιφέρει επιτέλου αυτή την σταθερότητα που τόσο έχει λύσει τα τελευταία 100 χρόνια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη δόκτωρα Καταρίνα Βόλτσικ. Ασχολείται στο Κέντρο για Ρωσικές, Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Μελέτες στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Ο κύριος Λούκας δεν θα είναι διαθέσιμος. Μόλις μας γνωστοποίησε ότι λόγω θανάτου του Χέλμουτ Σμιτ πρέπει να ασχοληθεί με τα εκδοτικά του καθήκοντα. Αυτά συμβαίνουν. Έχετε, τα... Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έξοχη εισαγωγή μου διευκολύνει τη ζωή, λέει η κυρία Βόλτσεκ. Ας σκεφτούμε την προσέγγιση της Ρωσίας όσον αφορά τους πολέμους διατυπωσόπων στην, στον εγγύς εξωτερικό της χώρο συνοψίζεται σαν πόλεμος με χαμηλό κόστος, χαμηλό κίνδυνο και με ωφέλη στατηγική. Εκ των πραγμάτων η κατάσταση περιεπλάκει αρκετά. Οποιοδήποτε πόλεμος αντιπροσώπων έχει εγγενείς κινδύνους που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε με μια επισκόπηση των πραγμάτων. Η Ρωσία χρησιμοποίησε θετικέ δυνάμει δύο φορέ. Στην Κρυμαία και στην, στο Ανατολικό Ντομπάσκ, στην Ουκρανία. Ε, και αυτέ οι δύο προσπάθειε συναθρίζονται, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικού σκοπού στην πραγματικότητα. Η Κρυμαία εμπεριέχει τρία στοιχεία. Έχουμε στοιχείο ποινή, τιμωρία, αποτροπή και πάνω απ' όλα αφορά την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Να διορθωθούν τα ιστορικά σφάλματα και η Κρυμαία είναι ένα μείγμα μεθόδων. Άρα είναι επιτυχές αποτέλεσμα ευρυδικού πολέμου. Είναι ένα κράμα επιχειρήσεων φανερών και μυστικών, πολύ προσεκτικά σταθμισμένων, ούτω ώστε να αποφευχθεί ή ε, ε, το να ξεπεράσει κανείς ε, την, το όριο που απαιτεί στρατιωτική απάντηση. Η Κρυμαία και εντός Ρωσίας και εκτός έγινε αντιληπτή σαν μια επιτυχία Ντομπάσκ. Το δεύτερο κομμάτι της σύγκρουσης είναι πολύ πιο περίπλοκη η περίπτωση. Η, πιο, η πλησιέστερη αναλογία είναι με άλλους παγωμένους πολέμους στην μετασοβιετική περιοχή. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι μια ψευδής αναλογία αυτή. Διαφορετικό στόχο, διαφορετικό χρονισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι παγωμένοι, οι παγωμένε συγκρούσει έγιναν αμέσω μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση και είχαν εθνοτική και εδαφική συνιστόσα σαφή και στον Ντομπάς αυτό λείπει. Αυτό που έχουμε στον Ντομπάς, χωρίς την εθνοτική συνιστόσα, έχουμε πάνω από 20 χρόνια που πέρασαν μετά την Σοβιετική Ένωση. Έναν πόλεμο διαντιπροσώπων που καλύπτεται σαν εμφύλιος πόλεμος. Κάτωθεν προσέγγιση, εξέσπασμα διαχωριστικών τάσεων που μεταμορφωθήκαν πολιτικώς σε δύο διαφορετικές δημοκρατίες λαϊκή δημοκρατία είναι η μήτρα που ε, έχει κληρονομηθεί από τη Σοβιετική Ένωση και χρησιμοποιείται στετική ισχύ σε πολύ περιορισμένο βαθμό για να επιτευχθούν, μάλλον να πιστούν. Είναι ένοπλη πυθός που χρησιμοποιείται. Η χώρα στόχος πίθεται να συμμορφωθεί με τα αιτήματα της δυνάμεως που παρεμβαίνει. στετική ισχύ χρησιμοποιείται μόνο στο βαθμό των αναγκαίων για να προωθηθούν πολιτικοί στόχοι και οι στόχοι θα έλεγα είναι του τουλάχιστον στο μετασοβιετικό χώρο. Πρόκειται περί διαχωρισμού ενός κομματιού της Ουκρανικής επικρατείας και να επανεισαχθεί αυτή η περιοχή υπό νέου πολιτικούς όρους που de facto θα δημιουργήσουν ένα είδος ρωσικού προτεκτοράτου ή θύλακα εντός μιας ενιαίας ενιαίου πολιτικού χώρου ουκρανικού. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο και επικίνδυνο σαν πολιτικός στόχος. Ε, γιατί αυτός ο στόχος. Κατά την άποψή μου, για να δημιουργηθεί μια νέου είδους εξάρτηση ε, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Πολλαπλές εξαρτήσεις έχει κληρονομήσει η Ουκρανία από τη Σοβιετική Ένωση. Εμπόριο, ενέργεια και πολιτική. Αυτά, αυτές οι εξαρτήσεις απέτυχαν όμως. Δεν έδωσαν στη Ρωσία την επιρροή που θεωρούσε σαν δεδομένη και που ανέμενε ε, στην γειτονική της περιοχή. Οπότε είναι ένας πολιτικός στόχος να δημιουργηθεί, να ξανασχεδιαστούν τα όρια και οι δομές του Ουκρανικού κράτους. Όμως αυτό ήταν επιτυχές μέχρι κάποιο όριο, διότι η Ουκρανία δεν έδρασε στη συνιστόσα αποτροπής έναντι των στατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας που είχαν συσσωρευτεί στα σύνορα την Ουκρανία. Είχα μια κλιμάκωση και αποκλιμάκωση στην Ουκρανία. Από υβριδικό πόλεμο που βασιζόταν σε μισθοφόρους και τοπικούς εθελοντίες κινηθήκαμε σε περιορισμένο πόλεμο που χρησιμοποιούνται μονάδες θετικές σε περιορισμένο βαθμό και για περιορισμένη χρονική περίοδο. Και αυτό μόνο για να διατηρηθεί η εικόνα εμφυλίου πολέμου η εντύπωση εμφυλίου πολέμου. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι για το ρωσικό κοινό που δεν θα μπορούσε να ανεχθεί το υψηλό κόστο τη παρέμβασης και μέχρι τώρα βλέποντα την αντίδραση στη Συρία μπορούμε να είμαστε πιο διστακτικοί για αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή για να πιστεί η Ουκρανία βασικά ότι πρόκειται περί εμφυλίου πολέμου άρα πρέπει η Ουκρανία να αναθεωρήσει τι περιφερειακέ δομέ για να συμπεριλάβει τον Ντομπά επί διαφορετική βάσεω. Διεθνώ όμω επιτρέπει επίση στη Ρωσία να αρνηθεί παρέμβαση, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία ή κάτι τέτοιο. Η Ρωσία μπορεί να εμφανιστεί σαν διαμεσολαβητής ειρηνευτικός. Αυτό διότι κατά κάποιο τρόπο η στρατηγική εξαρτάται σε περιορισμένη ισχύ και τελικά βασίζεται όμως στην Ουκρανία να δράσει συναρτήσει των πολιτικών ετοιμάτων. Γι' αυτό γίνεται κάτι ε, πολύ φιλόδοξο και άνευ προηγουμένου, αλλά και είναι μια στρατηγική που είναι παρακινδυνευμένη. Γιατί λέω ότι είναι παρακινδυνευμένη. Διότι η χρήση στατιωτικής ισχύω τελικά νομιμοποιεί τα αιτήματα της παρεμβαίνουσας δυνάμεως. Άρα χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη ισχύ και το είδαμε πριν την πρώτη συμφωνία του Μίνσκ και πριν τη δεύτερη συμφωνία του Μίνσκ. Είδαμε κλιμάκωση της ισχύω που νομιμοποιεί τα αιτήματα. Τι έχουμε τώρα όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Έχουμε ένα είδος αντίστασης. Δεν είδα ούτε ένα άτομο από την Ουκρανία που θα με τα χαρά στα εφάρμοζε τη συμφωνία 2 του Μίνσκ, τη δεύτερη συμφωνία του Μίνσκ και έχουμε τελικά μια αποτελμάτωση. Η συμφωνία η δεύτερη του Μίνσκ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ε, τι έχουμε στη διεθνή πρακτική κανονικά. Πρώτα μια συμφωνία καταπαύσεως του πυρός που ακολουθείται από πιο μακροχρόνια και λεπτομερέστερη πολιτική διευθέτηση μέσα στη σχετική συμφωνία. Η Μίνσκα 1 και 2, οι συμφωνίες, ε, δημιουργούν, ενοποιούν τις δύο διαδικασίες ένα. Και έχουμε από τη μία τη χρήση πολιτικής ισχύω με την πολιτική διευθέτηση από την άλλη και τα συγχωνεύουν. Μέχρι τώρα η σύγκρουση του Ντομπάς δεν έχει στόχο το πάγωμα, ούτε προσάρτηση αυτού του τμήματος της Ουκρανίας, πρόκειται περί αναθεωρήσεως των συνταγματικών δομών της Ουκρανίας και των στατικών δομών. Αυτό έχει κρατήσει πάνω από ένα χρόνο και μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι η πόλεμη είναι σχετικά φθηνή και η κατοχή είναι ακριβή. Και αυτό βλέπουμε στον Τομπάς. Η κλίμακα της κατοχής της ε, κατεχόμενης για την Ουκρανία της περιοχής αυτής είναι υψηλό το κόστος. Εκτιμάται περίπου στα 2,5 ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμα εκεί και η μισή από αυτούς είναι συνταξιούχοι οι οποίοι πληρώνονται σε ακατάστατα χρονικά διαστήματα και πρέπει να καλυφθούν. Και οι δημόσιες υπηρεσίες επίσης παρέχονται. επισκευάζονται ταχύτερα τώρα οι δρόμοι από ότι όταν ήταν υπεύθυνη η κυβέρνηση του Κιέβου για αυτή την περιοχή. Όμως αυξάνεται το κόστος και στα πλαίσια της γενικότερης ευρύτερης κρίσης δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκλειστεί. Μάλλον η ευρύτερη κρίση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό η παρεμβαίνουσα δύναμη είναι έτοιμη να εφαρμόσει θετική ισχύ ή να επιλέξει μια λιγότερο φιλόδοξη πολιτική διευθέτηση ίσως τελικά να μην εκπληρώνει τους στόχους της μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό για την Ουκρανία, για το θέμα αυτό και για τον ευρύτερο γενικότερο μετασοβιετικό χώρο είναι ότι μέχρι πέρσι πιστευόταν εκτενώς ότι υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ η Ρωσία μάλλον είχε δύο εξωτερικές πολιτικές. Μία για την εγγύης γειτονιά και μία για τον υπόλοιπο κόσμο. Εάν συγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική με ένα πληκτρολόγιο, είχαν δύο ξεχωριστά πληκτρολόγια οι Ρώσοι. Τώρα συγχωνεύτηκαν σε ένα πληκτρολόγιο που είχε περισσότερα πλήκτρα που χρησιμοποιεί για να παίζει τους στατηγικούς σκοπούς η Ρωσία. Οπότε ε, γίνεται πιο απρόβλεπτη η κατάσταση αλλά και ενδιαφέρουσα. Τελικά αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία εν συγκρίση με τις προηγούμενες εξελίξεις στην μετασοβιωτική περιοχή είναι ένα νέο μοντέλο ρωσικού στατιωτικού προβληματισμού που συνδυάζει παραδοσιακά στατιωτικά εργαλεία, αεροσκάφη και τάγκς που είναι αληθινά, στη Συρία Φερρυπίν, αλλά με νέα έμφαση που δίδεται στην έκπληξη, στοιχείο της έκπληξης, ε, στατηγικής και πώς ξεγελάς τον αντίπαλο. Και αυτό κάνει τα πράγματα απρόβλεπτα. Επίσης, από πλευρά τακτικής και τακτικών εξελίξεων σε σχέση με τους ευρύτερους πολιτικούς στόχους είναι ενδιαφέρον. Η βασική μου σύσταση θα ήταν όχι μόνο να εστιαστούμε επί των τακτικών εξελίξεων, αλλά να σκεφτούμε και τους ευρύτερους πολιτικούς στόχους που επιδιώκει η σε αυτή η δύναμη. Και εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσουμε τώρα την ε, συζήτηση. Σόλτ Νέμετα ναι, από την Ουγγαρία. Δεν έχει φτάσει ακόμα. another proxy Άλλος ένας πόλεμος για την προσώπων εδώ. Ο κύριος Ατσουμπάλης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε σαφείς ε, όταν κατονομάζουμε τα πράγματα. Να λέμε το πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι αντιπροσώπων στη γειτονιά μας είναι πόλεμοι εναντίον μας, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, ευρωατλαντικής ε, κουλτούρας. Αν δούμε την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, εύκολα εντοπίζουμε την επωνομαζόμενη ρωσική ευρωπαϊκή ατζέντα. Και αυτή η ατζέντα έχει αυτές τις προτεραιότητες. Να αναστείλει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιρροή της το, με το σοβιετικό χώρο. Να αποτρέψει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ενισχύσουν τον ρόλο τους. Να ενισχύσει ε, την οικονομική και ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Να ενισχύσει τους ε, υπέρμαχους και υποστηρικτές ε, του Πούτιν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να προάγει τις, τη διχόνοια και τις διαφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδυναμώσει γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η Ρωσία δεν αλλάζει και ο βομβαρδισμός ε, της Συρίας έχει οδηγήσει σε νέα κύματα μετανάστευσης από τη Συρία ε, προς τις γειτονικές χώρες και την Ευρώπη. Ακούμε επίσης ε, στοιχεία για τη νέα αρκτική οδό μετανάστευσης μέσω της Ρωσίας προς την Νορβηγία. Και οι Νορβηγοί αξιωματούχοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους για αυξανόμενες εισρωές μεταναστών, με τη στήριξη μάλιστα των Ρώσων. Αυτά είναι μερικά ορισμένα παραδείγματα της ρωσικής στρατηγικής αξιοποιώντας διάφορα μέσα για να κλιμακώσει την ε, επίθεσή της στην Ευρώπη και να επιβαρύνει τους ε, Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες καθώς πλησιάζει η στιγμή της αναθεώρησης των κυρώσεων προς τη Ρωσία ε, κυρώσεις που είχαν επιβληθεί ε, προς τη Ρωσία εξαιτίας ε, της προσάρτησης της Κρυμαίας. Ο αντίκτυπος των κυρώσεων και η απειλή νέων κυρώσεων είναι θεμελιώδης παράγοντας που απέτρεψε τον Πούτιν από το να συνεχίσει την επιθεσή του. Γι' αυτό θα πρέπει να εμείνουμε στους κανόνες μας και να τους ακολουθήσουμε. Είτε αυτό σημαίνει να καταπολεμήσουμε την πολιτική διαφθορά, να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια των πολιτικών μας κομμάτων ή να προβάλλουμε το όραμα της, ε, της Ευρώπης και να επισημάνουμε ότι βρίσκεται υπό επίθεση αυτό το όραμα. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου τώρα ο Πρόεδρος. Ο κύριος Πετρέα. Θα μιλήσω ρουμανικά. Ευχαριστώ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει πολύ αυτός ο πόλεμος στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνοι τους δεν μπορούν να σταματήσουν αυτή την κλιμάκωση. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε ε, την ε, συνεργασία μας και την εταιρική μας σχέση με το ΝΑΤΟ και θέλουμε να εξακολουθήσουμε να αποτελούμε γεωστρατηγική ενότητα και μονάδα στο μέλλον παρότι σε ό,τι αφορά την... Μιλούμε για την Μέση Ανατολή, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και ε, την, ε, τις άλλες παγωμένες, αν θέλετε, συγκρούσεις, την υπερδινιστερία και το καθεξής. Όλα αυτά δείχνουν την απειλή που υπάρχει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες που βρίσκονται στην ε, πλέον αδύναμη θέση σε ό,τι αφορά τους πολέμους προσώπων, ή είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της ε, ρωσικής και ουκρανικής ευρύτερης ε, γειτονιάς. η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση εισβολής της Ουκρανικής επικράτειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, πολύ μεγάλα σύνορα με αυτή τη χώρα. Προς το παρόν είναι ακόμα ασφαλή βέβαια αυτά τα σύνορα. Ευχαριστώ. Και να μιλούν οι συγητές που προηγήθηκαν δεν θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ποιος, ποιος είναι ο λόγος που γίνονται πόλεμοι και είναι οι περιελιστικές επεμβάσεις που γίνονται με στόχο τον έλεγχο των αγορών, τον έλεγχο του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, των δρόμων μεταφοράς τους. Αυτή είναι η ουσία. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση για αντιπροσώπους, εδώ υπάρχει η απόκρυψη ότι εκτός από τις, από τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις υπάρχουν και περιφερειακές και άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν τα δικά τους συμφέροντα και κάνουν πολέμους για τους δικούς τους λόγους και βεβαίως υπάρχουν κάθε αστική τάξη σε κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα, υπάρχουν μερίδες που ανταγωνίζονται, γι' αυτό λοιπόν δεν κάνει κανένας για την ψυχή της μάνας του, έχει συγκεκριμένη, ε, συγκεκριμένα συμφέροντα που τέμνονται και με μεγάλες δυνάμεις, γι' αυτό και γίνονται αυτοί οι πόλεμοι και υπάρχουν και οι ανταγωνισμοί. Επίσης, ε, θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Γιατί γίνονται ιστορικές αναφορές και διαστρεβλώσεις. Τι σχέση έχει άραγε ε, ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης και η βοήθεια στο Αφγανιστάν που ε, μπόρεσε και κατόρθωσε και υπάρχει για παράδειγμα έστω και για λίγο χρονικό διάστημα υπουργό Παιδείας γυναίκα. τα κορίτσια πήγαν στο σχολείο, υπήρξαν εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Τι σχέση έχει με τις Ναλπάλμ τη βαρβαρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Τι άφησε πίσω η Σοβιετική Ένωση με τα δικαιώματα αυτά που διακόπηκαν από τους Ταλιμπάν, το τέρας που εξέθρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες υπερελιστικές δυνάμεις, τι σχέση έχει με τη σημερινή κατάσταση και το χάλι μετά από δεκαετία, πάνω από δεκαετία υπερελιστική επέμβαση στο Αφγανιστάν, μόνο ναρκοφυτίες, φτώχεια και εκμετάλλευση και εξαθλίωση. Αυτός είναι ο κόσμος σας, αυτός ήταν ένας διαφορετικός κόσμος που ε, δεν ήξερα από εκμετάλλευση. Αυτή είναι η διαφορά, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στα ήδη υποθέντα από τους συναδέλφους. Αυτό που αποκαλούμε πόλεμους δια ε, αντιπροσώπων θα μπορούσαν να αποκληθούν και υβριδικοί πόλεμοι. Και υπάρχει και πολλή ε, τεκμηρίωση από αυτόν. Εμένα μου άρεσε η φιλανδική πρωτοβουλία πολύ. Πήραν μια ανάλυση, κάναν μια ανάλυση και μας έδωσαν και ένα φυλάδιο ε, στο Ελσίνκι όταν η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΣΑ έλαβε χώρα εκεί και το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι οι βρυδικοί πόλεμοι δεν είναι κάτι καινοφανές. Αυτός ο υβριδικός πόλεμος, αυτά τα υβριδικά στοιχεία υπήρχαν και κατά παρελθόν. Η Λιθουανία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Αν δείτε πώς έγινε η κατοχή μας το 1940, είχε υποθεί τότε ότι παρουσιάστηκε ότι είμαστε οι χαρούμενοι σαν χώρα, ότι συμφωνήσαμε να δεχτούμε αυτή την κατοχή. Αυτού του είδους οι πόλεμοι δεν είναι κάτι το καινούριο. Απαιτούν συντονισμό υψίστου επίπεδου. Υπάρχει ένα συντονισμός που απαιτείται μεταξύ των αρχών, των ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων. Και θα ήθελα να προσέξετε ε, το ρόλο που τα ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από τη Ρωσία παίζουν στη Δύση. Ξέρετε, μπορείτε να πάτε σε κάποια δυτική χώρα, να ανάψει την τηλεόρασή σου σε αυτή τη χώρα, στο ξενοδοχείο και να ακούσει σε τέλεια αγγλικά. Υπάρχει τηλεπτικό κανάλι που λέγεται Russia Today, δεν ξέρω να αλλάξω όνομα, το Russia Today τέλο πάντων. Ακούτε το κανάλι και αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι αυτά που λένε είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τι ΗΠΑ και τίποτα χειρότερο από τη Δύση. Και το σκέφτομαι αυτό. Αν ο κόσμο τα ακούει αυτά τα πράγματα, αυτή την πλήση εγκεφάλου, τη δέχεται καθημερινά, που παρουσιάζεται σε άπτε στα αγγλικά, βέβαια γίνεται πλήση εγκεφάλου επιτυχή. Και μπορούμε να αισθανθούμε την προπαγανδιστική αυτή μηχανή της Ρωσίας ε, που ακούγεται στους εθέρες. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί για να εμποδίσουμε οι κοινωνίες μας να παραπλανηθούν από αυτό. Διότι ο πόλεμος πρόκειται να ξεκινήσει. Αυτή είναι η τελευταία φάση της προετοιμασίας για τον πόλεμο. Τώρα η βασική μάχη θα είναι για τα μυαλά και τις καρδιές των λαών και δεν θα πρέπει να χάσουμε σε αυτόν τον τελευταίο πόλεμο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αντίθετα από ό,τι ελέγχθη προηγουμένως, έχουμε μαζί μας τον Edward Lucas από το Λονδίνο. Είναι ε, από τους ε, εξέχοντες συντάκτες του, του Economist και πολιτικός αναλυτής επίσης. Ευχαριστούμε που είσαι παρόν, έστω και εξ και θα ήθελα να σου ζητήσω να λάβεις το λόγο για 10 λεπτά. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να μπορέσω να σας μιλήσω με βιντεοδιάσκεψη. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πέθανε μόλις ο Χέλμουντ Σμίτ, όπως ξέρετε, και έγραφα την νεκρολογία του, η οποία θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα του Economist. Σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αν μπορώ λοιπόν να παρουσιάσω τον εαυτό μου, Αντιμετωπίζω τα θέματα αυτά εδώ και πολλά χρόνια, παρακολουθώ τα ζητήματα της Σοβιετικής Ένωσης από την εποχή του ψυχρού πολέμου και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι προσπάθειες των αντιφρονούντων ήδη από την εποχή του σιδηρού παραπετάσματος και με ενδιαφέρουν τα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας ακόμα και όταν ορισμένοι θεωρούν ότι έχουν επιληθεί όλα αυτά τα προβλήματα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πρόσφατα, μάλλον όχι ακριβώς πρόσφατα, το 1994 στο Αμβούργο εδώ μια ομιλία ο Helmut Σμιτ και προειδοποίησε για τις δυνατότητες, τις πιθανότητες να προέλθει κάποια επίθεση από την πλευρά της Ρωσίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ακόμα και όταν οι περισσότεροι κόσμοι, άνθρωποι δεν έδιναν καμιά σημασία να σκεφτούμε αυτό το θέμα και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι είχαν δίκιο. Οι Αστονοί, οι Λιθουανοί, οι Λετονοί, οι Τσέχοι κτλ. Όλοι αυτοί οι οποίοι ε, ανησυχούσαν για θέματα τα οποία εκείνη την εποχή η Δύση τα είχε αφήσει κατά μέρο, σαν να μην ήταν σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να ακούμε τις απόψεις αυτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως τα έλεγα, αυτό το οποίο είπε ε, ο Λιθουανός συνάδελφος γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν μια ουσιαστικά εχθρική και ακόμα και σχεδόν πολεμική ε, στάση της ε, Ρωσίας εναντίον τους. Η έννοια του πολέμου δι' αντιπροσώπου είναι πολύ εύστοχη. Είναι η χρήση κάποιου άλλου για να κάνει ένα πόλεμο ε, προ όφελό του και χρησιμοποιούν ένα αντιπρόσωπο για να έχουν τη δυνατότητα διαψευσιμότητος. Εάν τα πράγματα πάνε στράφη, α, όχι δεν το κάναμε εμεί, το κάνει κάποιο άλλο. Ο βουλευτή από την Ελλάδα που έλαβε το λόγο προηγουμένω είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα υπεριαλισμού. Ναι, φυσικά. Και αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του, του ψυχρού πολέμου είχαμε πολέμους διαντιπροσώπων και από την πλευρά των Σοβιετικών και από την πλευρά των Αμερικανών. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυτικό κατά κάποιο τρόπο ή ιδιαίτερα ρωσικό σε σχέση με τη χρήση αυτών των τεχνικών. Αν μιλάμε όμως για εμπεριαλισμό θα πρέπει να προσέξουμε να μην μπερδέψουμε τις ειδικέ συνιστώσεις. Είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για στην Αφρική και στην Ασία, αλλά και η Ανατολική Ευρώπη έχει υποστεί τον υπεριαλισμό της Σοβιετικής Ένωσης και εξακολουθεί να τον υφίσταται σε κάποιο βαθμό. Αν κάποιος λοιπόν ενδιαφέρεται ως αριστερός για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το τι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία και τι μπορεί να συμβεί και στα βαλτικά, στις βαλτικές δημοκρατίες στη συνέχεια. Εμείς στη Δύση αγωνιζόμαστε για να δούμε τι προσπαθεί να κάνει η Ρωσία με αυτού του πολέμου διατυπωσόπων Γιατί προσπαθούμε να κατηγορηποιούμε τα πράγματα. Λέμε αυτό είναι θέμα αστυνομικό, αυτό είναι θέμα μυστικών υπηρεσιών, αυτό έχει να κάνει με ενέργεια, αυτό έχει να κάνει με εισαγωγέ και εξαγωγέ, έχει να κάνει με το επιχειρήν. Είναι θέμα βασανιστήριων κτλ. Όλα τα βάζουμε σε κουτάκια. Έχουμε ειδικού φορείς, έχουμε θεσμικούς φορείς, έχουμε την επαγγελματική η ηθική που ακολουθούμε για να ταξινομήσουμε τις διάφορες αυτές τις ενέργειες. Αλλά ίσως αυτός που είναι απέναντί μας δεν έχει αυτές τις νοητικές κατηγορίες στο μυαλό του. Μπορεί να κάνει κάποιος προπαγάνδα το πρωί, να ασχολείται με συλλογή πληροφοριών το μεσημέρι, να ασχολείται με τα θέματα ενέργειας το απόγευμα και το βράδυ με τα θέματα διαφθοράς. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία συντονισμένη σειρά ενεργειών από τη Ρωσία, γιατί αυτό έχει να κάνει με την δομή της ε, ε, Ρωσίας που Γίνονται αυτές οι προσπάθειες μέσω της Gazprom, μέσω των hackers οι οποίοι επιτίθενται στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιώντας τη δύναμη της διπλωματίας, τη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας, την ικανότητά της να κάνει προπαγάνδα. Όλα αυτά όμως είναι παράλληλες ενέργειες και πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και Εμεί δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Λέμε, αν είναι ενεργειακό θέμα θα πρέπει ο ρυθμιστής ενέργεια να επιληφθεί. Αν είναι προπαγάνδα, κάποιο άλλο. Εκεί επιτυγχάνει πιστεύω η Ρωσία, γιατί θέλω να τονίσω ότι η Ρωσία μέχρι στιγμή κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Εμεί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι γίνεται. Εμεί ουσιαστικά δεν θέλαμε να ακούσουμε, δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα. Η Ρωσία έχει κάνει σημαντικές πρόοδους έχει καταφέρει να φέρει τα βρώμικα χρήματα μέσα στην πολιτική, έχει εξασφαλίσει τη δημιουργία οικονομικά εξαρτημένων κρατών, έχει σημαντικά ενισχύσει την στρατιωτική της ικανότητα. Στη δεκαετία του 90 η στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας ήταν ένα ανέκδοτο, δεν μπορούσε να κάνει περίπου τίποτα. Τα τελευταία 15 χρόνια όμως έχει τροποποιηθεί αυτή η κατάσταση. Έχουν λοιπόν σημαντικές ικανότητες, έχουν πυράβλους κρούς που μπορούν να ε, φτάσουν από την Κασπία τη Συρία, έχουν πολύ καλό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα, έχουν πολύ καλές ειδικέ δυνάμεις, έχουν πολύ καλή συλλογή πληροφοριών, έχουν ε, προχωρημένα, εξελιγμένα όπλα. Η Ρωσία λοιπόν προχωρεί και προχωρεί επίσης και σε επίπεδο προπαγάνδας. Πριν από 20 χρόνια δεν θεωρούσαμε ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με την ρωσική προπαγάνδα. Όχι. Θεωρούσαμε το 1991 ότι η Ρωσία θα έχει ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης, θα πήγαν όλα τα πράγματα μια χαρά και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά ο, η Ρωσία έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει μια γυαλιστερή και επιτυχημένη μηχανή προπαγάνδας η οποία μπορεί σιγά σιγά να παραμορφώνει την αλήθεια. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε πάντα αυτά τα οποία μπορεί να λέγονται από ένα επίσημο φορέα. Η Ρωσία όχι. Η Ρωσία όχι. Και αυτά φαίνονται όχι μονάχα στον, ε, στον τηλεοπτικό φορέα το RT, αλλά και σε άλλες ε, πολλές φορές ε, στα δικά μας μέσα ενημέρωσης που παίρνουν, στο διαφημίσει που παίρνουν πληρωμένες διαφημίσεις από τη Ρωσία που φαίνονται ότι είναι απλώς πληροφοριακού χαρακτήρα για τη Ρωσία, αλλά τις συγγράφουν αυτές τις διαφημίσεις πληρωμένοι ε, ε αξιωματούχοι που πληρώνονται από το Κρεμλίνο για να το κάνουν αυτό. Βλέπουμε λοιπόν και τις επιπτώσεις όλης αυτής της ε, προσπάθεια στον τομέα τη ενέργειας. Βλέπουμε τα αποτελέσματα στη Λιθουανία του τρέτου ενεργειακού πακέτου και το πώς η Gazprom προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, να εμποδίσει οποιαδήποτε προσπάθεια πραγματικής διαφοροποίησης ε, πηγών προμήθειας. Για να το εμποδίσει αυτό, τους δίνει μια μεγάλη έκπτωση για να το κάνει αυτό. Και με την Πολωνία πάλι. θα υπάρξει μια αντίστοιχη κατάσταση. Λοιπόν, ε, μάλλον η, Ρωσία, η Πολωνία έχει προχωρήσει γιατί έχει σταθμό συλλογή φυσικού αερίου που τη δίνει κάποια αυτονομία. Έχουμε πετύχει κάτι, αλλά τα πράγματα προχωρούν. Θυμάστε την κυβερνοεπίθεση το 2007 κατά της Εστονίας, τον πόλεμο του 2008 κατά της ε, ε, Γεωργίας. Χρησιμοποίησαν ε, διακομιστές που ήταν έξω από τη Ρωσία για να χτυπήσουν την Εστονία, ώστε κανείς να μην μπορεί να τους κατηγορήσει. Η επίθεση κατά της ε, Γεωργίας ξεκίνησε από την Απχαζία και πάλι ήταν αντιπρόσωποι της ε, Ρωσίας η επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Ντονέσ και τον Λουχάνσκ που ουσιαστικά ήταν δορυφόροι της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν έχει αποκτήσει μια μεγάλη πείρα στα θέματα αυτά και εγώ είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Αν συμφωνείτε καλό είναι, αλλά θα ήθελα να ακούσω ε, θέσεις αντίθετες, οι οποίες θα με κολλήσουν στον τοίχο ενδεχομένως. Ευχαριστώ. Thank you very much. I hear that you will still... Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσετε τη συζήτηση και θα απαντήσετε και σε τυχόν ερωτήσεις. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Τσόλτ Νέμετ από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ, Ελμάρ. Και καλωσορίζω και, τους, ε, και τον συνάδελφο Εντ Lucas. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερα εμπιστευμένη αυτή ανάλυση. Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο παράλληλους πολέμους. Και εξετάζουμε ξεχωριστά αυτούς τους δύο πολέμους. Εγώ θα ήθελα να σε συγχαρώ, Ελμαρ. Ή μάλλον να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να τους εξετάσουμε από κοινού. Γιατί έχουμε πόλεμο στη Συρία και έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι ίσονος σημασίας το ερώτημα της ε, σύνδεσης των δύο ζητημάτων, γιατί συνδέονται. Δεν είναι τυχαίο που εν μέσω του πολέμου Ουκρανίας και Ρωσίας βρέθηκαν ρωσικά αεροσκάφη στη Συρία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και πρέπει να εξετάσουμε τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πολέμων. Και τώρα έχει συσταθεί η διαδικασία της Βιέννης. Είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην διαδικασία της Βιέννης και το Ιράν και η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Αλλά με την άλλη διαδικασία τι γίνεται. δίνεται η απαραίτητη προσοχή από την διεθνή κοινότητα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει αντίστοιχη προσπάθεια, διαδικασία επίλυσης του ουκρανικού ζητήματος. Αν όχι, θα πρέπει τουλάχιστον στο νου μας να έχουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική επίλυση. Και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Θα ήθελα κι εγώ να αναφέρω αυτό που είπε ο Λούκας, ότι πρέπει να ακούμε τους φίλους μας ε, στην πρώτη γραμμή, στις χώρες της πρώτης γραμμής. Τα ιστορικά τους αντανακλαστικά είναι πολύ ωφέλιμα και πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Ίσως και αυτή είναι τους Κορυφής ε, να του ΝΑΤΟ μάλλον, ε, θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και η διάσκεψη της Βαρσοβίας. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη μελλοντική πολιτική επίλυση της ε, ρωσο-ουκρανικής ε, σύγκρουσης, θα πρέπει να έχουμε κάποιες αρχές κατά νου. Ίσως η πιο σημαντική από αυτές, μια κόκκινη γραμμή θα έλεγα, είναι ότι οι κατεχόμενες χώρες όπως η Γεωργία, η Ουκρανία δεν θα πρέπει να βρεθούν στην κατάσταση όπου να μην είναι σε θέση να έχουν και να διατηρήσουν την αυτοκυριαρχία τους και να, ε, την αυτοδιάθεσή τους και να προσδιορίσουν το μέλλον τους. Κάποιες φορές χρειάζονται πολιτικές συμφωνίες, όμως αυτή είναι μια γραμμή την οποία δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε η εθνική κυριαρχία της Γεωργίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συναντηθήκαμε, Edward. Καλώς ήρθες στην Επιτροπή. Το δέχομαι ότι η θετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και η προσάρτηση της Κρυμαίας είναι απαράδεκτα γεγονότα. Καταδικαστέα, τα έχω καταδικάσει επανειλημμένα εκ μέρους ομάδας μου στην Επιτροπή. Και βέβαια οι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν μπορούν να έρθουν ενώ Ουκρανική επικράτεια είναι τελή υπορωσική κατοχή. Και συμφωνώ με την ανάλυση σου για το ρόλο τη Ρωσία σήμερα και του καναλιού Russia Today. Ε, μου ζήτησαν συνέντευξη και δεν την παρουσίασα τη συνέντευξη διότι επέκρινα αυτά που συμβαίνουν στο Κρεμλίνο. Και η διαφθορά των πολιτικών κομμάτων. Ακούμε το εθνικό μέτωπο της Γαλλίας ε, που υπερασπίζεται τα ρωσικά συμφέροντα σε αυτή την επιτροπή παρόλο που από ό,τι καταλαβαίνω τους έχουν δανείσει ε, ρωσικές τράπεζες, μάλλον τράπεζες με ρωσικά χρήματα, τους έχουν δώσει χρήματα στο Παρίσι. Λοιπόν, ε, ο εχθρός του εχθρού τελικά γίνεται φίλος σου. Και ξέρω ότι κατά παρελθόν εσύ και εγώ συζητήσαμε την υποστήριξή σου για τους Τσετσένους στον πόλεμο κατά της Μόσχας εδώ και 10 χρόνια παρόλο που τώρα που μόνο που επιστρέψα από το Κουρδιστάν οι τρομοκράτες Τσετσένοι θεωρούνται ότι είναι οι χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι και πολεμούν για το Ισλαμικό κράτος και σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέτωπα όπως είναι Αζερβαϊτζάν κατά Αρμενίας για τον Αγκόρνο Καραμπάχ πρέπει να πω ότι υποστηρίζω τη ρωσική εμπλοκή που υπερασπίζεται τους Αρμένιους τη θέση τους για το Ναγκόνο Καραμπάχ εναντί των Αζέρων και στη Συρία Μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακός ο Ασάτ, τον υποστηρίζουν το Ιράν και η Ρωσία και ε, υποστηρίζουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι και η Σαουδική Αραβία την αντιπολίτευση παρόλο που τελικά πηγαίνουν όπλα σε φοβερές τυχαντιστικές ομάδες και ίσως και το ίδιο το Ισλαμικό κράτος. Η εξωτερική πολιτική είναι πάντα πολύ περίπλοκη και πολύ θεαζώνη προσπαθώντας να καταλάβει κανείς ποια είναι τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να αποσυνδέσουμε τη θέση μας στη Δύση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική και σύμμαχοι έναντι των όσων έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία ή ποια είναι η απειλή που αντιπροσωπεύει έναντι των βαλτικών χωρών από αυτά που ίσως να κάνει στον Κάφκασο η Ρωσία, αυτά που προσπαθεί να κάνει στη Συρία η Ρωσία. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με του Ρώσου, να του ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει όλοι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με του Ιρανούς, του Σαουδάραβε, του Τούρκου, του Αμερικανού και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε την κατάσταση στη Συρία. Διότι σαφώ ο εμφύλιο πόλεμο στην Συρία με αυτή την έξοδο των πληθυσμών και τη ροή ε, των μεταναστών δημιουργεί υπαρξιακό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εγχείρημα και πρέπει να κάνουμε εξισορρόπηση διλημάτων. Ποια είναι τα συμφέροντα σε ένα μέτωπο και να τα συγκρίνουμε αυτά τα συμφέροντα με αυτά που έχουμε σε ένα άλλο μέτωπο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Έντουαρτ για αυτά που είπες και τη συμβολή σου σε αυτή την ουσιαστική συζήτηση. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα Κατά τη δική μου άποψη, κανένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον πόλεμο πληροφοριών ή τους υβριδικούς πολέμους, τουλάχιστον όπως τα βλέπουμε τώρα τα πράγματα. Είμαι πεπισμένος κι εγώ ότι η Ρωσία κάνει πραγματικά ένα πόλεμο πληροφοριών εναντίον μας, παρά το γεγονός ότι δεν το έχουμε αναγνωρίσει στην πλήρη κλίμακα του φαινομένου. Ένα παράδειγμα η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων έχει δημιουργήσει μια ειδική μονάδα για την Ανατολική Ευρώπη που έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους ε, εταίρους μας ε, στην Ανατολική Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν το, την πλημμυρίδα πληροφοριών που έρχεται από τη Ρωσία στις χώρες αυτές. Χρειαζόμαστε όμως και μια West Stratcom, αντίστοιχη της East Stratcom, που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη μας να υποστηρίξουν σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο την αντιμετώπιση αυτών των στοιχείων προπαγάνδας και να εξηγήσουμε στον λαό μας τι είδους παραπληροφόρηση προσπαθούν να φέρουν σε εμάς οι Ρώσοι. Τα μηνύματα αυτά είναι πράγματι τρομακτικά. Ένα παράδειγμα στην Ουκρανία έχουν διαδώσει ότι ένα νεαρό αγόρι σταυρώθηκε στο Ντονέτσκ. Στο έδαφος το οποίο ελέγχεται από την Ουκρανική κυβέρνηση. Το κάναν τόσο ωραία ώστε ο κόσμος σοκαρίστηκε από αυτά τα νέα. Βρήκανε κάποιον ο οποίος είπε ότι το είδε και εξήγησε πολύ λεπτομεριακά τι έγινε. Αλλά οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί είπαν όχι αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν πολύ αργά γιατί η είδηση είχε περάσει σε όλο τον κόσμο ήδη. Είχε μείνει στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Η δυτικοί λοιπόν δημοσιογράφοι έχουν κάποια όρια τα οποία δεν ξεπερνούν ποτέ. Αλλά δεν υπάρχουν ποτέ τέτοια όρια στην, ε, στα μυαλά των Ρώσιων και προσπαθούν να μας πρόξουν, να μας βάλουν στη γωνιά. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε αντισταθεί με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή μας, ενώ αυξάνεται η πίεση από τη ρωσική πλευρά. Η έκκλησή μου είναι λοιπόν όπως λέει ο Έντουαρτ και άλλοι εμπειρογνώμονες, ότι θα πρέπει να πούμε στους πολιτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ ότι είναι απαραίτητο να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τη ρωσική προπαγάνδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο πόλεμος δια την δεν γεννήθηκε σήμερα, αλλά εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Πιστεύω όμως ότι η επέκτασή του και η δημοφιλία του εδράζεται επί της αρχής της ευθύνης των μεγάλων χωρών και στόχο έχει τη δημιουργία φόβου. Αν δεν υπήρχαν τα πυρηνικά οπλοστάσια, πιθανότατα ήδη θα είχαμε άλλον ένα παγκόσμιο πόλεμο, όπως είπε κάποιος. Είναι αυτά συνέπεια, αυτά τα γεγονότα είναι συνέπεια που δημιουργούνται από δύο στοιχεία. Το πρώτο, η κρίση εκείνων των χωρών που σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα ουσιαστικά ε, διαλύονται και αυτές είναι οι, ρίζες των συγκρούσεων. Και δεύτερο στοιχείο που είναι στο επίκεντρο του πρώτου είναι από τον, ε, την αποστολική προσέγγιση που ακολουθούν για, εκδημοκρατισμό η ΕΠΑ. Σαν να του έχει ανατεθεί στη ΣΥΠΑ αυτός ο ρόλος ε, μετά το 89. Το ρώτημά μου. Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα ισορροπία Πολλοί πιστεύουν ότι στην Ανατολική Ευρώπη ο μόνος δρόμος είναι να αποφευθεί ο υποχρεωτικός προσιλητισμός και να δημιουργούνται ε, ουδέτερες χώρες ε, που είναι σαν ε, διαχωριστικό φράγμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται μια πολιτική με βάση την ισορροπία των δυνάμεων. Νέα ισορροπία δυνάμεων καρπός νέας γεωπολιτικής που δημιουργήθηκε από αυτά τα γεγονότα. Άλλοι πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να θέσουμε τροχοπέδι στις ορέξεις της Ρωσίας από την περίπτωση αλλά και άλλων χωρών είναι να δώσουμε νέο πρωταγωνισμό, πρωταγωνιστικό ρόλο μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Υπάρχει κάποια δυσκολία εκεί όμως. Χρειάζεται ρητή συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ακόμα διαιρέσει εντός μας. Ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω και εγώ μερικέ παρατηρήσει. Και μετά καταληκτικά θα ζητήσω από τους καλεσμένου μα να δώσουν μια απάντηση σε ερωτήματα που τέθηκαν. Είπε ο κύριος Λούκας ότι με την αντιμετωπίσει της Ρωσίας. Η Ρωσία φαίνεται να κερδίζει την αντιπαράθεση. Εγώ πιστεύω ότι έχει δίκιο στο θέμα αυτό. Πάντα ένα αυταρχικό καθεστώς έχει μεγαλύτερη ευκολία να αναπτύξει μια στρατηγική που συνενώνει όλες τις συνιστώσεις από ότι μια δημοκρατία. Η δημοκρατία ζει σε μια πολυμορφία, υπάρχει διαφορά μεταξύ πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εξουσίας και υπάρχουν πολλές αλληλοσυγκρόμενες τάσεις. Αλλά η ιστορία μας δείχνει ότι οι δημοκρατίες σε τελική ανάλυση πάντα κερδίζουν οι αγώνες για την ελευθερία, πάντα μπορούν να κερδίσουν και ιδίως όταν έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει μια δημοκρατία, ένα δικτατορικό, ένα αυταρχικό καθεστώς. Η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Χωρίς τώρα να υπάρχει κάποια, ε, κάποιος παραλληλισμός η η Μεγάλη Βρετανία φαινόταν το 40 να είναι τελευταία ζωντανή δημοκρατία στην Ευρώπη και φαινόταν απελπιστική η κατάστασή της. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κερδίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν εμείς να σκεφτούμε ότι αυτά πρέπει να είναι τα πραγματικά θεμέλια της δημοκρατίας που πρέπει να διατηρηθούν. Οι αυταρχικές εξουσίες μπορούν να αποφασίζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από την μακροσκελή διαδικασία που ακολουθούν τα κοινοβούλια μας, αλλά αυτό το πλεονέκτημα που τους δίνει τελικά δεν μπορεί να αντέξει στη μεγαλύτερη δύναμη που έχει η δημοκρατία. Δίνω το λόγο στην κυρία Βόλτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές οι απόψεις αποκούστηκαν μερικά σχόλια από πλευράς μου. Νομίζω ότι ένα στοιχείο ήταν ο πόλεμος κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνώ από αυτού ότι η Συμφωνία Σύνδεσης είναι η πρώτη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου από ό,τι γνωρίζω που έχει οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόκληση ανεπροηγούμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου είναι κάτι το οποίο γίνεται παντού ανά τον κόσμο και ιδίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται κατά κόρον. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι οι εμπορικέ σχέσει έχουν και πλέον και μια διάσταση ασφαλεία. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο. Είναι κάτι λοιπόν με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, αλλά και η αντίληψη των υπολείπων για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ε, την προαγωγή της δημοκρατίας ή του εμπορικού τους μοντέλου, που από πολλούς θεωρείται ε, παρέμβαση, παρεμβατισμός κ.ο.κ. Επομένως πρέπει να δούμε τον, τους νέους τρόπους ε, οικοδόμησης δεσμών μεταξύ υπήρων και χωρών. Αλλά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει απορροφηθεί ότι η ενσωμάτωση και προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας, ε, μια απειλή για την ασφάλεια των χωρών της μετασοβιετικής ε, περιοχής ε, που δεν θα πρόκειται, από την οποία δεν πρόκειται να επιβιώσουν. Εγώ ήμουν τώρα στο Αζερβαϊτζάν είναι από τι πλέον ε, ανεξάρτητες χώρες ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική τη. και η συζήτηση ήταν για τη σχέση μεταξύ Ρωσία και Αζερβαϊτζάν. Επομένω, έχουν αποδεχθεί τον ηγετικό, ηγεμονικό μάλλον ρόλο της Ρωσίας σε αυτόν τον χώρο και το μοναδικό στοιχείο είναι η ετοιμότητα ανάπτυξης στρατιωτική δύναμη. Επομένω, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Πώ δηλαδή οι ενέργειε άλλου παίκτη, άλλου φορέα δηλαδή, ε, επηρεάζουν και την αντίληψη που έχουν οι τρίτοι για την ε, πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν αξιοποιηθεί και καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Όμως, έχουμε ξεχάσει όλα αυτά τα μαθήματα που είχαμε αντιλήσει στο παρελθόν, γιατί νομίζαμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Είχα συνομιλήσει με μία αξιωματούχο ε, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και την είχα ρωτήσει για τον Ιβρυδικό πόλεμο και αν έχει κάνει κάτι το Ηνωμένο Βασίλειο από αυτού. Και μου είπε, ξέραμε ότι έπρεπε κάτι να κάνουμε, γιατί ήταν αυτή η Ιβρυδική πόλεμη πάντα στην ατζέντα μας, αλλά πάντα υπήρχαν πιο επίγοντα ζητήματα. Και έτσι από στρατηγική σκοπιά ε, στην Κρυμαία βρεθήκαμε όπτου» το οποίο βεβαίως ήταν ιδιαίτερα υπολογισμένο ε, και σωστά ενορχιστρωμένο, ούτως από την άλλη πλευρά, ούτως ώστε αυτά τα στρατιωτικά μέσα να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή. Το τελευταίο, ήταν, ή μάλλον πρώτο τελευταίο, αφορά την ε, Συρία και την Ουκρανία. Η Συρία και η Ουκρανία διαφέρουν, αλλά έχουν και ομοιότητες. Οι ομοιότητες είναι ότι ε, κάνουν ε, παρουσιάζουν την Ρωσία ως βασικό παράγοντα επίλυσης ε, της κρίσης για τη Δύση. Δεν πρέπει να υπάρξει δηλαδή λύση χωρίς τη Ρωσία μέσα. Και ταυτόχρονα αυτό συνδέεται και με την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί για να επιληθεί η κρίση της Κρυμαίας προς όφελος της Ρωσίας. Υπάρχει λοιπόν διασύνδεση των δύο, ότι δηλαδή πλησιάζει περισσότερο η Ρωσία προς την πλευρά ε, της δύση. όμως το τελευταίο και πιο σημαντικό είναι μακροπρόθεσμη, βράχη πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασυμβατότητα μεταξύ δύο στοιχείων. Θέλουμε την αδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας και την εθνική κυριαρχία χωρών όπως η Ουκρανία για παράδειγμα που τους επιτρέπει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πρέπει να δούμε πού θα μπει η κόκκινη γραμμή. Εάν η συμφωνία του Μίνσκ υλοποιηθεί με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται από τη ρωσική πλευρά, τότε θα είχε σταματήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης ε, της, ε, και προσέγγισης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όμως ε, μια θέση που δεν δημιουργεί ε, πραγματικά τακτικά ε, προνόμια για μια θέση που έχει πολύ μεγάλες ζημίες και θυσίες. Ευχαριστώ. Ερχόμενος από τις ΗΠΑ, εξεπλάγει να το πώς εδώ το Κοινοβούλιο ναι, έχει αντιληφθεί το τι γίνεται στη Ρωσία. Είναι διαφορετικά αυτά που ακούω εδώ σε σχέση με αυτά που λένε στη Ουάσιγκτον. Μέχρι Έχουμε νέο πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, δεν θα γίνει τίποτα διαφορετικό στη Ουάσιγκτον και δεν θα πρέπει να περιμένετε πολύ βοήθεια από την ε, Ουάσιγκτον. Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω, όντα αισιόδοξο, είναι ότι οι διατυπωσόπων πόλεμοι είναι καλοί αν μπορούσε να του χρησιμοποιεί σωστά, οι υβριδικοί πόλεμοι. Πάμε σε αυτό που είπα για το ασύμετρο κόστο. Για κάθε δολάρι που δαπανεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΙΠΑ δαπανούν σε αυτού του πολέμου πρέπει να ξοδέψει η Ρωσία χίλια δολάρια και σε κάποια φάση τελικά θα πονέσει. Και έτσι πρέπει κανείς να παίξει το παιχνίδι. Και όσο εμπλέκονται σε περισσότερες συγκρούσεις και μέτωπα οι Ρώσοι με περισσότερους πόρους που απαιτούνται, τόσο ψηλότερο το κόστος για αυτούς. Και η αντίστροφη όψη του νομίσματος είναι ότι αν τιμέ της ενέργειας παραμείνουν χαμηλέ και αν υπάρχουν πολλές άλλες πηγές ενέργειας πέρα τη Ρωσία, τα έσοδα θα μείνουν σταθερά και μακροπρόθεσμα η Ρωσία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν αυτό είναι ο στόχο. Δεν θέλω να είμαι πολύ κοινικό, θέλω να ρεαλιστή, είναι και το ανθρώπινο κόστος για τους ανθρώπους, τους ντόπιου ε, μέσω για τους πολέμους αντιπροσώπων. Και ο ανθρώπινο παράγοντας έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κύματο των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και από το Λίβανο κλπ. Αν δούμε τα οικονομικά μοντέλα τη ε, κρίσεω των προσφύγων. Και αν παίξει κανεί τα χαρτιά του σωστά υπάρχει ένα τρόπο να αντιστρέψει αυτό για αύξηση του ΑΕΠ τη περιοχή όταν εγκατασταθούν αυτοί οι πληθυσμοί. Πολιτικό είναι δύσκολο να γίνει γιατί είναι αλλοδαπή, διαφορετική θυσία, διαφορετικέ ζωέ κλπ. Οικονομικό όμω είναι εργατικά χέρια. Κάποια εργατικά χέρια είναι καλά εκπαιδευμένα έχουν δεξιότητε, επιχειρηματίε ε, και με τα χαρά θα δημιουργούσαν ανάπτυξη, θέσει απασχόληση, ε, επιχειρήσει. Ξέρω τη Συρία πάρα πολύ καλά, κυρίω του Σύριου και θα μπορούσε να αυξηθεί το ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, μέσω της μόχλευσης λόγω των προσφύγων που έρχονται από το Λεβάντε που τελικά θα κάνουν πιο ισχυρή την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποδυναμωθούν οι αντίπαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λουκ. Λούκα. Uh, Για τον Charles Τάνοκ πρώτα απ' όλα. ο ψυχρός πόλεμος ήταν πάρα πολύ μπερδεμένο. Πολλές φορές υποστηρίζαμε καθεστώτα και άτομα τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα και ελκυστικά με την ελπίδα ότι τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίζαμε τους κομμουνιστές που θεωρούσαμε πολύ χειρότερους. Ο ψυχρός πόλεμος στην Ευρώπη ήταν πολύ πιο απλός. Εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη αν με ενοχλούν περισσότερο οι Κινέζοι κομμουνιστές για αυτά που έκαναν στο Θιβέτ έναντι αυτών που κάναν οι Ρώσοι στην Τσετσενία. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ουδέτερα σαν άσκηση, σαν παραδείγματα της άσκησης πολιτικής δύναμης. Όταν πρόκειται για τους συμμάχους μας και τους φίλους μας, για τις χώρες που θέλουν να είναι σαν και εμάς, εκεί πρέπει να τους υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς και τις άλλες χώρες και φυσικά τις χώρες που είναι ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Αζερμπαϊζάν εναντίον της, ε, εναντί της Αρμενίας τα πράγματα είναι πολύ πιο ε, πολύπλοκα. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι η αιτία της τρομοκρατίας από την Τσετσενία οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισαν στη δεκαετία του 1990. Για το θέμα των στρατηγικών επικοινωνίων και του τρόπου να το κάνει η Δύση, συμφωνώ απόλυτα. Το, η δεξαμενή σκέψη στην οποία εργάζομαι στι ΗΠΑ είπα, έχει πολλέ ιστορίε ανθρώπων που έχουν άμεση εμπειρία στα κράτη της πρώτης γραμμής, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες τους να την φέρουμε την εμπειρία στις πρωτεύουσες της Δύσης, να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους λήπτες αποφάσεων για τα μέσα ενημέρωση, τους εκδότες και τους δημοσιογράφους, για να μην αφήσουμε να κάνουν κατάχαση της πληροφορίας οι Ρώσοι. Είναι γεγονός ότι οι δυτικοί δημοσιογράφοι είναι εκπαιδευμένοι να δίνουν αξία στην ισοδίκαια παρουσίαση των απόψεων. Ενώ από την πλευρά της Ρωσίας δεν ισχύει αυτό. Λένε, ξέρω εγώ, ότι το αεροπλάνο το οποίο της Μαλαισιακής, ε, Μαλαισιακών αερογραμμών, το MH17, ότι το ρίξανε οι ίδιοι Ουκρανοί. Αλλά αυτά είναι ουσιαστικά σαν τη διάκριση μεταξύ αστρονομίας και αστρολογίας. Αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν και δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουν. Πράγματι, θα πρέπει να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα Υπάρχουν πολλές φορές χώρες με ευγενείς ιδέες, ελεύθερες χώρες οι οποίες έχουν συντριβεί από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Σκεφτείτε χώρες όπως η Βρετική Δημοκρατία. Χώρες που είχαν θεσμούς που ε, καταστράφηκαν και άλλους που νομίζαμε ότι οι θεσμοί τους θα τους οδηγούσαν σε μεγάλες δυσκολίες αλλά τελικά επεκράτησαν. Νομίζω ότι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η Ρωσία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούν να κερδίσουν κάποιες νίκες. Έχω κάθε ελπίδα λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε, αλλά δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί και να παναπαυόμαστε, αν θέλουμε να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λέει και ο Πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συζήτησαν μαζί μας Έχουμε εστιάσει πολύ στην Ρωσία και στην ε, ανατολική μας γειτονία, αλλά έχουμε συζητήσει και για την ε, Μέση Ανατολή και την νότια γειτονιά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ασχοληθήκαμε με το θέμα των πολέμων δια αντιπροσώπων και τις περιπτώσεις του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας που αγωνίζονται για την τοπική και περιφερειακή επικυριαρχία στην περιοχή τους. Στην Ανατολική Ευρώπη τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα πίσω από τις κουρτίνες, να δούμε τι γίνεται στα παρασκήνια και επομένως να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και να διαμορφώνουμε τις κατάλληλες στρατηγικές. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε συμφωνίες οι οποίες μας αποδυναμώνουν παρά τα φαινομενικά τους πλεονεκτήματα. Αυτό ισχύει λοιπόν με την, στην περίπτωση της Ρωσίας η οποία ήδη έχει εμπλακεί και στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Δεν πρέπει να, ε, να παραδώσουμε τα όπλα στην περίπτωση της Ουκρανίας λοιπόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το πούμε με σαφήνεια ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε λανθασμένες κατευθύνσεις, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ο, στη Ρωσία ότι και αυτή έχει κάθε συμφέρον να, αγωνιστεί κατά της ε, τρομοκρατίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει και μουσουλμανικός πληθυσμός στη Ρωσία και που μπορεί να υπάρξει ε, αρνητικός αντίκτυπος στη Ρωσία από αυτά. Μας ενδιαφέρει όμως και να εξασφαλίσουμε ότι χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία και η Ουκρανία δεν θα απειλούνται από την Ρωσία. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ και θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήταν παρόντες σήμερα. Νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ έντονη σειρά συζητήσεων από χθε το απόγευμα μέχρι σήμερα και εγώ βρήκα πάρα πολύ και καρποφόρες αυτές τις ε, συζητήσεις και ιδίως το γεγονός ότι συμμετέσχανε και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτές τις ε, συζητήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε εδώ και σε άλλους χώρους να συνεχίσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Καλό ταξίδι επιστροφής ή καλό βράδυ στις Βρυξέλλες έχει πολλά μειονεκτήματα στη πόλη των Βρυξελών, αλλά κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κουζίνα των Βρυξελών. Σας εύχομαι λοιπόν ένα καλό βράδυ ή στις αιστείες σας ή στις Βρυξέλλες, τέλος της συνεδρίας σας